Okay, we will make a start. Um, we've just been told, uh, Mrs. Θα ξεκινήσουμε γιατί η συγγήτρια θα έρθει σε λίγο. Committee agenda this afternoon is the adoption of the agenda. Second. Μήνυμα από του διερμηνείς. Βρισκόμαστε στην 21η ημέρα των κινητοποιήσεων και δεν έχουμε δει καμία αντίδραση από την πλευρά τη διοίκηση. Αντίθετα σκληραίνει τη στάση του Γενικού Γραμματέα, Πολλές καμπίνες έχουν επιταχθεί και ω ένδειξη αλληλεγγύη δεν θα προβεί η ελληνική καμπίνα σε στάση εργασία, Απλά θα διακόψουμε ακριβώ στην προγραμματισμένη ώρα λήξης συνεδρίας. Ευχαριστούμε. Uh, uh, Ευχαριστούμε για τη δήλωση. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της μερισσίας διάταξης, που είναι η δημόσια ακρόαση για τις κρατικές βοήθειες και τη γνώση και χρηματοδότηση. Θα ξέρετε, πριν από κάποιο καιρό, είχαμε μια μελέτη για τις κανόνες περικρατικών ενισχύσεων, έρχεται και ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή η συγγήτρια. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια μελέτη για τους κανόνες περιγρατικών ενισχύσεων και καλό είναι να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα Έχουμε την εισηγήτρια. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ, να ευχαριστήσω και για την παρουσία εδώ του ομιλητέ μα. Από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι κρατικέ σχέσει και σχετικοί κανόνε ε, δεν είναι πάντοτε οι σωστοί. Στην περίπτωση του Brexit, ε, στην προλογική εκστρατεία, ε, όταν το ερώτηση τι αλλαγέ θέλετε να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί έλεγαν ότι δεν του άρεσαν κανόνε περί κρατικών ενισχύσεων. Αλλά εμεί που καταλαβαίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την ευθύνη γι' αυτό, έπρεπε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι κανόνε αντίθετα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουμε κανόνε για να το πετύχουμε αυτό και να μην υπάρχει στρέβλωση τη αγορά. Ε, γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων. Βέβαια. Σίγουρα δεν είναι δημοφιλής σε πολλού και γιατί δεν του καταλαβαίνουν ίσω πολύ και εκεί είναι ένα πρόβλημα και σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει μια επιφύλαξη απέναντι στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και μια επιφυλακτικότητα, διστακτικότητα ε, να γίνει υποδεκτό ένα σχήμα χρηματοδότηση που μπορεί να μην είναι σύμμορφο με αυτού του κανόνε. Όμω, οι μικρομεσαίε επιχείρησει ιδίω και οι μεγαλύτερε ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, για αυτού του κανόνες. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώ μια μικρή εταιρεία δεν μπορεί άμεσα να αποφεληθεί από την ουσιακή χρηματοδότηση. Πολλά λοιπόν αυτά που γίνονται. Σίγουρα είναι δύσκολο να κατανοήσουν όλες τι λεπτομέρειε. και έτσι ε, απλουστεύουν τα πράγματα και λένε ότι δεν είναι καλή αυτή η κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Σήμερα θα συζητήσουμε όλα αυτά και γι' αυτό οργανώσαμε την ακρόαση σήμερα. Είναι και η συγγήτρια εδώ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Θα τη δώσω το λόγο. Ινές, να κάνεις εσύ πρώτα τις αγωγικές παρατήρησεις και θα περάσουμε στο πάνελ των ειδοκών μας μετά. Ε, Αγιά Σέντερ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Ντέρεκ. Πάρα πολύ δίκιο είχες σε αυτά που είπες και στην Επιτροπή μας. Μας απασχόλησε αρχικά το πώς ε, θα επεξεργαστούμε αυτό το θέμα προϋπολογισμός, έλεγχος εφαρμογής ε, και εκτέλεση προϋπολογισμού και τα τελευταία χρόνια έδειξε ξεκάθαρα η πολύπλοκευτή κατάσταση ότι υπάρχει διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για ιστορικούς λόγους. Ε, είχαμε τα ταμεία της επιχορηγήσης που ε, διακλαδώθηκαν με άλλα χρηματοδοτικά μέσα με το blending τώρα που έχουμε, καταλήγουμε να έχουμε σχέδια μέσω μακροπρόθεσμα, πολύπλοκα έργα. Εγώ ασχολούμαι στην Επιτροπή με τα, πολυ... με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά υπάρχουν και άλλα με μεγάλες εμβέλειες μακρόπνοα έργα, όπω ε, έχουμε δίσοντα με τον υποδομών. Και η ανάγκη που δημιουργείται είναι να υπάρξει μια διαφοροποίηση, μια διάκριση ώστε με τρόπο συνεκτικό να μπορούν τα έργα αυτά να λάβουν ε, κάποιες ε, μορφές ενίσχυσης. Να είναι επιλέξιμα για να πάρουν κάποια ενίσχυση. Και επίση έρχεται να υπάρχει μια προσθετικότητα. Ε, έχουμε την σηματοδοτημένη, αλλά να υπάρχει και μια ξεκάθαρη προσθετικότητα και δέσμευση, όλο και σαφέστερη δέσμευση μέσα των κρατών μελών για αυτά τα μεσοπλάσμα μακροπρόθεσμα έργα. Να είναι δηλαδή ξεκάθαρο αυτή η δέσμευση να μην δίνεται, ε, να μην γίνεται κατά περίπτωση και ότι κάθε φορά κυβέρνηση να αλλάζουν και τα πράγματα, αλλά να έχει ξεκινήσει σημαντικέ επενδύσεις να συνεχίζονται. Και στην Επιτροπή μας ε, αυτό μας απασχολεί. Οι δεσμεύσεις αυτές, οι επενδύσεις αυτές Ιδίω έργα υποδομών που υπάρχει μεγάλη ε, συνιστόσα ανταγωνιστικότητας. Και μιλάω για τομείς που πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε που πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες περί ενισχύσεων και με ποιο τρόπο οι ανάδοχοι, οι δικαιούχοι και οι διάφοροι άλλοι φορείς που θα συμμετέχουν στην χρηματοδότηση των έργων θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Και όλοι οι συμμετέχοντες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε κάποιες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ακριβώς για να ξεκαθαριστεί ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στον τομέα της απλούστευσης και της εφαρμογής των ε, κανόνων να είναι πιο απλοί οι κανόνες και πιο ξεκάθαρη η εφαρμογή τους για να μην τίθεται υποπίεση ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της μελλοντικής χρηματοδότησης για συγκεκριμένα έργα και πολιτικές ευρωπαϊκές. Εξού λοιπόν και θεωρήσαμε ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε εδώ αυτή την ακρόαση, να μας εξηγήσει η Κομισιόν τι γίνεται. Πρόσφατα είχαμε κάποιες εξελίξεις. Και βέβαια στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προπολογισμό και όλες τις ε, επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, καλό θεωρήσαμε ότι θα ήταν να έχουμε αυτή την ακρόαση για να διαφωτιστούμε σε ό,τι αφορά τις διατάξεις αυτές, την εφαρμογή των κανόνων στη δικαιούχη και η ανάδοχη των έργων να έχουν ξεκάθαρη ιδέα. Πού είναι σαφείς και υποχρεωτικοί οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και πού αντίθετα χρειάζεται και εκεί θα δώσουμε την έμφαση από πλευρά της δική μας Επιτροπής στις επενδύσεις και στον προπολογισμό. ώστε να είναι καλύτερα, ώστε το δυνατόν πιο ε, μεγάλη αξιοποίησή του, του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού. Ελπίζω λοιπόν να είναι καλή ακρόαση. Εύχομαι κάθε επιτυχία τις εργασίες και θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που μας ε, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα, τα πολύπλοκα ζητήματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην πρώτη συζήτηση. Στο πρώτο τμήμα, πώς παρακολουθεί τη συμμόρφωση ε, των κρατών μελών με του περικρατικών ενισχύσεων κομισιών. Έχουμε τέσσερι ομιλητέ. Κύριο ε, Κούκμαν είναι ο πρώτο ε, στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κοντ. It's a real pleasure to be here this afternoon. Uh Apologies. Um, to, uh... Μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Να σας πω πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα στην ε, Κομισιόν. Είμαι υπεύθυνο γι' αυτό στην Κομισιόν και γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα προσωπικά. Για να ξεκινήσω, ε, νομίζω είναι καλό να υπογραμμίσω τους στόχους που ο Πρόεδρος σύντομα παρουσίασε, ότι δηλαδή να εξασφαλίσουμε πως οι κρατικές ενισχύσεις μέσω της χρήσης δημοσίων πόρων δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. και δεν εκδιώχνουν τις επενδύσεις ιδιωτών. Να εξασφαλίσουμε πως είναι ε, συστατικό της εσωτερικής αγοράς που δεν ε, όμως ρευλώνει τη λειτουργία της. Επίσης είναι σημαντικό να μην δίνονται κρατικές ενισχύσεις στους παραγωγούς ώστε να έχουν ε, τη δίκαιες ευκαιρίες να κερδίσουν ένα μερίδιο της αγοράς. Και τέλος είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε πως εκεί όπου παρεμβαίνουν τα κρατημέλη μέσω της χρήσης των ε, δημοσίων πόρων ε, συμβάλλουν στην οικονομική ε, ευημερία και την ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εντεταγμένο στην συνθήκη, καταγεγραμμένο στη συνθήκη και άρα είναι μία από τις παλαιότερες κοινοτικέ πολιτικές. Όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, σημαίνει πως οι κρατικές ενισχύσεις απαιτούν τα κράτη-μέλη στην χορήγηση δημόσια, κρατικής ενίσχυσης να μπορούν να καλύψουν γενικές, ε, γενικά προβλήματα της αγοράς, δηλαδή να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει στόχος κοινού ωφέλειας, δεν μπορεί να δίνονται χρήματα έτσι. Δεύτερον, θα πρέπει να περιορίζονται τα χρήματα, Δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική αποζημίωση, ε, δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν δε τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις ε, που είναι ευθές ε, σε κάθε περίπτωση και δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τη λειτουργία της, να βλάπτουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε να διατηρήσουμε την οικονομική ειρήνη στην εσωτερική αγορά και να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότητά της. Δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και την, τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ξέρουμε ακριβώς γιατί τι πράγμα μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή, ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία εφαρμόζονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεσα από τον προπολογισμό, δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις και άρα δεν υπόκειται στους ελέγχους για κρατικές ενισχύσεις. Όλες οι άμεσες παρεμβάσεις όπως το Horizon, το, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, όλα τα χρήματα προέρχονται άμεσα από τον προπολογισμό και τα οποία διαχειρίζεται η Ένωση η ίδια, είναι εκτός του πεδίου ελέγχου των ε, κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε τούτου λεχθέντος και ο Λιβιέ που κάθε δίπλα μου θα πει περισσότερα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την συνοχή με την τις πολιτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρούνται ε, ότι πρέπει να υπόκεινται στους ε, ελέγχους περικρατικών ενισχύσεων. Αντίθετα, τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, εκεί που τα χρήματα, τα χρήματα δίνονται στα κρατημέλη, ώστε τα κρατημέλη να τα διαχειριστούν σε ευρεία, ευρεία προβλή, ε, project, αυτά υπόκεινται στους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Αυτή η διάκριση νομίζω είναι σημαντική ε, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Όταν λοιπόν αυτό το εφαρμόσουμε βλέπουμε ότι μόνο 10 με 20% όλων των δαπανών υπό τα Ευρωπαϊκά Διαρθωτικά Ταμεία υπόκεινται στον ε, έλεγχο περικρατικών ενισχύσεων. Το μεγαλύτερο τμήμα των διευθυντικών ταμείων δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Δεύτερον, η Κομισιόν ως τμήμα μιας ε, απλοποίησης και εξυγχρονισμού έχει εξαιρέσει συνολικά το μεγαλύτερο μέρος του μικρού τμήματος που μένει για, ως κρατική ενίσχυση. Τι σημαίνει αυτό, ότι σύμφωνα με πολύ απλούς κανόνες που μπορούν να εφαρμόσουν και τα ίδια τα κατημέλη μόνα τους, τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται πλέον να κοινοποιούν προς την ε, Κομισιόν την κρατική ενίσχυση πριν την καταβάλουν, αλλά μπορούν αμέσως να ε, συνεχίσουν με τα προγράμματά τους ε, απλά σε επόμενους κανόνες. 10 με 20% όλων των δαπανών λοιπόν είναι κρατικές ενισχύσεις και μόνο το 10% εξ αυτού, δηλαδή 1 με 2% πρέπει να κοινοποιείται προς την Επιτροπή εξάντε εκ των προτέρων. Στην πράξη δηλαδή είναι ελάχιστα τα project που πρέπει να κοινοποιούνται και να εγκρίνονται. Και αυτά τα project τα οποία κοινοποιούνται, δηλαδή το 1 με 2% στην πράξη, στην πραγματικότητα, ε, δεν θέτουν δυσκολίες και πολύ γρήγορα εγκρίνονται μάλιστα. Πρόκειται για τεράστια προγράμματα, πολύ σημαντικά, αλλά παίρνει περίπου 5 μήνες για να τα εγκρίνουμε. Ε, βέβαια, ε, ακούγεται, γίνονται πολλές συζητήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις ε, και για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Όμως είναι σημαντικό να δούμε και τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι ότι πολύ μικρό κομμάτι των κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνεται στο ΕΣΥΦ, δηλαδή στο σχέδιο Juncker, στο ΕΤΣΕ, στα ελληνικά. ωστόσο είναι α, σαφές ότι εξασφάλιση της εφαρμογής και της στήριση των κανόνων είναι πολύ σημαντικό. Ε, να γίνεται και επίσης είναι πολύ σημαντικό να, ελέγχονται αυτό, να ελέγχεται αυτό το μικρό ποσοστό κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να ελέγχεται. Γι' αυτό και έχουμε πολύ εργαστές σχέση με τους συναδέλφους στην DG Radio ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτάχυνση τη εξέταση όλων αυτών των στοιχείων και έχουμε φτιάξει και ένα κοινό σχέδιο δράση ώστε να ε, ε, υπάρξει μεγαλύτερη κοινοποίηση των όσων ισχύουν στα κράτη-μέλη. Μας ανησυχεί, είναι σημαντικό και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι διευκολύνει τη ζωή των υπαλλήλων στα κράτη-μέλη που πρέπει να δαπανίσουν τα χρήματα. Γιατί θέλουμε να δαπανηθούν τα χρήματα σωστά, αλλά και γρήγορα. Είναι σωστό λοιπόν να πει κανείς ότι ε, τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ε, μπορούμε να, τα όσα μπορούμε να μετρήσουμε είναι ενθαρρυντικά σχετικά. Τα στοιχεία για λάθη στους ελέγχους, που είναι αντικειμενική παράμετρος, δείχνουν πολύ σημαντική μείωση των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια. Και, κατά συνέπεια, το κομμάτι των, του σφάλματος ως ποσοστό συνολικό φαρμακευτικού όγκου φάρματος είναι εξαιρετικά μικρό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω που θα πρέπει να μας ενθαρρύνει. Ήδη εν συντομία μίλησα για τις την τον ευρύ εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των βελτιώσεων, πιστεύω, και είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε αυτήν την ε, ε περικοπή που μίλησε, για την οποία μίλησε και η συγκήτρια. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων που ε, βαραίνουν πια ως ευθύνες τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμως η Κομισιόν εργάζεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να διευκολύνει την ανάληψη ευθύνης από πλευράς τους. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη σειρά διαδικασιών πέρα από τις ε, εταιρικέ σχέσεις στις οποίες ήδη ανεφέρθηκα. Να σας δείξω, δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε μια ομάδα εργασίας με τα κατημέλη που όπου μοιραζόμαστε καλές πρακτικές γιατί τελικά την ευθύνη φέρουν τα κατημέλη και μπορούν να μάθουν. Είμαι ένα από τους ΔΕ και προσπαθούμε αυτό να το διευκολύνουμε. Έχουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για να βοηθήσουμε να ε, λυθούν ε, ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Υπάρχει πολύ εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης και επισκέψεων στα Εγώ επισκέπτομαι τα κρατη όλα τα κράτη-μέλη ε, και οι συνάδελφοί μου και υπάρχει μεγάλο μερίδιο υλικού κατάρτισης με κεντρικά σημεία συντονισμού σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί σε κάθε κράτος μέλος είναι η καρδιά της γνώσης όσον αφορά την ε, νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και μπορούν να ενημερώνουν και να βοηθήσουν τις, αρχι... τις αρχές ε, ανα πάσα στιγμή. Έχουμε ένα συνάδελφο εδώ που ήταν υπεύθυνο για τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων στην Πολωνία. Η κεντρική μονάδα ε, ε, ε, συντονισμού στην Ελλάδα επίσης έχουμε έναν εκπρόσωπο εδώ, έχουμε το Συμβούλιο Ανταγωνισμού στη Ρουμανία που έχει αυτή την ευθύνη και υπάρχει και μια μονάδα στη Γερμανία στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων που είναι υπεύθυνο. Αυτή η σημαντική λοιπόν συνεργασία με τα κέντρα συντονισμού σε κάθε χώρα. Ως τμήμα Συγγνώμη, αλλά ήδη κλείσατε τα, τελειώσατε τα 10 σας λεπτά, τα εξαντλήσατε. Εντάξει, να σταματήσω. Αλλά νομίζω πως αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα... δεν θα χρειαστεί ο χρόνος αυτός ε, για τους συναδέλφους. Εντάξει, τότε θα τον αφαιρέσω από εκείνους, λέει ο Πρόεδρος. Ως τμήμα λοιπόν αυτής της προσπάθειας έχουμε εξετάσει με τα κάτι μελη για να δούμε τι προκαλεί τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των διορθωτικών ταμείων. Και δεν είναι ένα εμπειρικό σύνολο ποσοτικών στοιχείων, δεν είναι άποψή μας, είναι η άποψη των ανθρώπων που εργάζονται για αυτά τα θέματα. Και όπως μπορείτε να δείτε από τις πιθανές αιτίες, τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η περιπλοκότητα, ο περίπλοκος χαρακτήρας των ίδιων των διευθυντικών ταμείων. Και Επίσης, κάποια άλλα χαρακτηριστικά του ρυθμιστικού πλαισίου που δεν είναι δηλαδή κρατικές ενισχύσεις οι ίδιες ε, πρώτο στοιχείο δυσκολίας είναι πέμπτο ή έκτο στον κατάλογο. Ε, όταν ζητάμε, ρωτάμε από τα κάτι μέλη τι πιστεύουν ότι είναι η, ε, το πρόβλημα, θα σας πούνε ότι οι κρατικές ενισχύσεις παίζουν ένα σχετικά περιορισμένο ρόλο. Αυτό βέβαια στηρίζεται και από την διάρκεια και την ταχύτητα που ανέφερα, όπου μπορούμε να δούμε ότι Εάν συγκρίνουμε το σύνολο εξαιρέσεων και τα μέτρα τα οποία κοινοποιούνται και δείτε πόσο γρήγορα μπορούν να εφαρμοστούν, θα δείτε ότι ο ροζ στήλη που είναι το κομμάτι της συγχρηματοδότησης, θεωρητικά κατά μέσο όρο εφαρμόζεται σε 1,5 μήνα. Σε αντίθεση με την μη συγχρηματοδοτούμενη κρατική ενίσχυση που παίρνει περίπου 3 μήνες μέχρι ότου εφαρμοστεί. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και θέλουμε βεβαίως να συνεργαστούμε με τα κατημέλη για να το βελτιώσουμε και άλλο. Και κλείνω λέγοντας ότι για το μέλλον έχουμε φιλοδοξίες να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα και σε αυτό το πλαίσιο ότι στο πλαίσιο του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα θέλαμε να ευθυγραμμίσουμε ακόμα περισσότερο τις κρατικέ ενισχύσεις και τους σχετικούς κανόνες όπου τα κρατικά χρήματα συνδυάζονται με τα ευρωπαϊκά. Για παράδειγμα, έτσι ώστε οι κανόνες να εντάσσονται με τρόπο ώστε να συνδυάζονται χωρίς πρόβλημα και να ε, εκτελούνται πιο γρήγορα. Και οι συνάδελφοί θα πούνε κάποια περισσότερα θέματα. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και βέβαια για την αριστεία, που είναι ένα πραγματικό πρόγραμμα έρευνας, αλλά και για όσα μέτρα εμπίπτουν στις συνολικές εξαιρέσεις, που θέλουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω. Η κατάσταση βελτιώνεται. Από τις πληροφορίες που έχουμε φαίνεται ότι ε, βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά σίγουρα θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία σας και για την ε, παρέμβασή σας ε, και να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, ο κ. Βάλμπρακ, ο οποίος είναι επικεφαλής από τη Γενική Διεύθυνση Budget. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και Νομίζω ότι είναι λογικό το ότι συζητάμε για τους κανόνες ε, ε, της Ευρωπαϊκής χρηματοδότηση και κοιτάμε λοιπόν το κείμενο αυτό το πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και η Επιτροπή μας σας ξέρει γνωρίζει καλά το κείμενο αυτό και ξέρουμε ότι στις 23 Ιουλίου θα τεθεί εφαρμογή μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο, η οποία αναμένεται και από την, μετά την έγκριση και από το Συμβούλιο. Να αναφερθώ λοιπόν στους νέους κανόνες, γιατί νομίζω καλύτερα είναι να συζητάμε το μέλλον και το πώς θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες αυτοί. Τι βρίσκουμε λοιπόν σε αυτόν τον χρήκο τον κανονισμό. Δεν γίνονται πολλές αναφορές σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τους απλούς λόγους τους οποίους ε, ήδη ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή στην άμεση διαχείριση τέτοια ε, κρατική ενίσχυση όταν οι πόροι εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συνεκτικότητα λοιπόν αναφέρεται σε έναν τομέα της ε, χρηματοδοτικές εγγύησης και ο, εκεί βρίσκουμε τις ίδιες αρχές τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως. Πρέπει να επιλύσουμε φυσικά προβλήματα και αποτυχίες της αγοράς, να κοιτάξουμε το θέμα συμπληρωματικότητας, να δούμε τις επενδύσεις από όλες τις πηγές, να υποστηρίξουμε οικονομικά βιώσιμους ε, και να κοιτάξουμε και τη σύνθεση και να είμαστε φυσικά και συνεκτικοί σε ό,τι αφορά την ε, συνοχή με τους ε, κανόνες ε, των κρατικών επιδοτήσεων. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ κοντά στην αγορά, όντω. Από την άλλη, συνήθω είμαστε σε έμεση διαχείριση, όχι σε άμεση διαχείριση. και η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις αρχές ε, του ελάχιστου μετόχου. Αυτό δεν ε, ισχύει μόνο για την χρηματοδότηση και τις εγγύησεις. Και έτσι εφαρμόζονται λοιπόν οι ίδιες αρχές ε, ό,τι αφορά τις εγγύησεις ε. και σε ό,τι αφορά τις ε, επιδοτήσεις. Αν υπάρχει δηλαδή υποστήριξη των επιδοτήσεων με το οικονομικό μέσο, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, μια εταιρεία να παρουσιάσει ένα έργο, να το χρηματοδοτήσει με τα μέσα, με τις χρηματοδοτικές εγγυήσεις, θα καλυφθεί αυτό και από τις ίδιες αρχές. Άρα το όλο ζήτημα είναι ευρύτερο από ότι το, υπό τη έννοια. Ένα σημαντικό στοιχείο. Η αξιολόγηση. Το παράδειγμα το οποίο δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επεξηγηματικό σημείο μας σε ό,τι αφορά τον νέο χρηματονομικό κανονισμό ανέφερε το εξής. Ο στόχος είναι να αγγιθούμε αξιοπιστία από μία αρχή, από μία υπηρεσία όπου αυτό είναι δυνατόν. Και αναφέρεται λοιπόν αυτή η αρχή της ε, συμβατότητας, της συνοχής. Έχει λεχθεί λοιπόν αυτή η συνεκτικότητα για τις κρατικές ενισχύσεις. και οι οικονομικοί παράγοντες θα πρέπει να εξαρτώνται από την έγκριση αυτή που χορηγείται και φυσικά δεν θα πρέπει να αλλάζουν οι κανόνες. Αυτό φυσικά είναι κάτι ευαίσθητο. Και θα το δούμε αυτό και σε λίγο όταν οι συνάδελφοι αναφερθούν ε, στα όσα ισχύουν για τα δεύτερη ταμεία. Ύστερα υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ισχύει σε ό,τι αφορά την έμεση διαχείριση. Όταν θα επιλεχθεί λοιπόν ο ενδιάμεσος, αυτό θα πρέπει να γίνει με ετυλογημένο τρόπο, εκ των προσδέρων, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπό φυσιολογικέ συνθήκε. εργαζόμαστε με την ΕΤΕΠ αλλά και με τις εθνικές τράπεζες ε, πρόθεσης. Αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει ένα ευαίσθητο σημείο σε ό,τι αφορά και τη γενικότερη πτυχή του ανταγωνισμού. Αυτές αρχές λοιπόν που δεν έχουν αλλάξει, πώς έχουν αποτυπωθεί στα καινούργια προγράμματα για το μέλλον, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση στο μέλλον. Αυτό θα εξετάσουμε τώρα, στην ε, συντομία. Έχουμε δύο βασικά παραδείγματα τα οποία ήδη έχουν αναφερθεί από τον κύριο Κουκάν. Το ενιαίο, την ενιαία ομάδα κανόνων και την ε, σφραγιδαριστία σε ενιαία ομάδα κανόνων σημαίνει ότι όλοι οι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί στο μέλλον θα κρατήφονται άπαξα. Ε. Πάντα με αναφορά στον χρηματοοικονομικό κανονισμό για την ε, συμβατότητα με, την κρατική, με τις κρατικές ενισχύσεις, τις κρατικές και σε ό,τι αφορά τον ε, ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση. Θα απλοποιήσει την ζωή και των ε, ενδιαμέσων και των εταίρων δηλαδή, αλλά και των δικαιούχων. Θα υπάρχει μία συμφωνία με κάθε κυβέρνηση και με τους ε, φορείς που εφαρμόζουν τα προγράμματα. Μία συμφωνία αντιπροσωπεία, μία ενιαία θηρίδα για όλη την εφαρμογή των εργαλείων αυτών. Και τα κράτη-μέλη δεν θα χρειάζεται να κοινοποιούν εκ νέου την, Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκ νέου χορήγηση χρηματοδότησης εφόσον φυσικά δεν αλλάξουν οι όρικοι συνθήκε τη παρέμβαση. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η σφραγίδα αριστεία. Την ανέφερε και ο κύριο Κούκαν. Δηλαδή, αν κάποια προγράμματα έχουν ε, ελεγχθεί σε επίπεδο ορίζοντα 2020 και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης πόρων, μπορεί να χρηματοδοτηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκών ε, κρατών μελών βάσει του ESF+, του EFRD και το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα LIFE. Άρα δεν χρειάζεται εκ νέου αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα του προγράμματος. Και δεν χρειάζεται λοιπόν να λεχθεί πάλι συμβατότητα με τους κανόνες για τους, ε, τις ευρωπαϊκές ε, διτάξεις. Θα πρέπει λοιπόν συνοψίζοντας ε, να δώσουμε σημασία σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα και τη συνοχή των κανόνων και για προγράμματα τα οποία περνούν από κεντρική διαχείριση, όπως είναι το Connecting Europe, ε, Connecting Europe Facility, ορίζοντας 2020. Θα δείτε στο, στα εκτιμώντες αυτής της νέας πράξης διάφορες αναφορές σε ό,τι αφορά την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση της οικονομικής πλευράς και σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ε, που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Η κυρία Φερνάνδες Ούτς τώρα από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. rules apply to an increasing share of cohesion policy spending. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, πολιτική συνοχή για την περίοδο 2020, εστιάζεται στην ανάπτυξη, στι θέσει απασχόληση και τι επενδύσει. Και ω εκ τούτου σημαντικά ποσά συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα, για παράδειγμα ευρυφάσμα, ενέργεια και ανεώσιμε ενέργειε και η υποστόρεξη των οικονομικών δραστηριοτήτων ε, μπορεί να χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Η κρατική ενίσχυση τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ε, ως ένα σημαντικό, μια σημαντική πηγή σφαλμάτων από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ωστόσο, ο αριθμός των σφαλμάτων αυτών έχει μειωθεί το περσινό έτος από 20% το 2014 σε μη ποσοτικοποιημένα ποσοστό σφάλματων το 2016. Ο βασικός ε, λόγος ε, για τα σφάλματα αυτά ήταν η εσφαλμένη ερμηνεία των κανόνων ε, ελληπίκης κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλήματα σε ό,τι αφορά την επιλογή των προγραμμάτων για συγχρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχει κάνει για να μειώσει λοιπόν το ποσοστό σφαλμάτων αυτό. Καταρχάς, ε, ο κοινός κανονισμός διατάξεων για την περίοδο 2020 έδωσε διατάξεις για αρισιμότητα εξάντα, προκειμένου να υπάρχει σωστή επένδυση. Ένας από τους όρους αυτούς λοιπόν έχει να κάνει να υπάρχουν διατάξεις για την εφαρμογή κανόνων σε ό,τι αφορά τους πόρους αυτούς. Ε, και αυτό σημαίνει ότι εντολή, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντολή να ζητήσει διευκρινήσει ε, από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που επιμένουν οι αδυναμίε. Στην αρχή τη προγραμματική περίοδου, πέντε κράτη-μέλη δεν τήρησαν αυτέ τι διατάξει εξάντε. Πλέον όλα τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται. Όπω είπε και ο κ. υπήρχε ένα σχέδιο δράση το οποίο εγκρίθηκε το 2015 και το οποίο θα εξεταστεί εκ νέου τώρα το 2018 σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και έγινε ένας εξυγχρονισμός και μια απλοποιηποίηση του πακέτου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το σχέδιο δράσης ε, περιλαμβάνει ένα σκέλο σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση που χορηγείται προ τα κράτη-μέλη και κατά δεύτερον ένα σκέλο εκπαίδευση. Ε, έχουμε, για παράδειγμα, εκπαίδευση για τους ελεγκτές, ε, για άλλους φορείς κρατικούς υπάρχουν και στρατηγικές, ε, στρατηγική εκπαίδευση για κάποιους τομείς, ανατομέα δηλαδή, και για τους εμπρεκνόμονες σε, σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. Και μεγάλο τμήμα βασίζεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ανταλλαγές μεταξύ ομοτήμων, ε, στρογγυλές τράπεζες, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπου ανταλλάσσονται οι εμπειρίες και τελικά καταρτίζονται κάποια έγγραφα τα οποία βρίσκουν σύμφωνο όλους τους συμμετέχοντες και επίσης άμεση ενίσχυση και εργαλεία άμεσης ενίσχυσης για την υποστήριξη δήμων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης. Η συνεργασία μεταξύ της DigiComp και της DigiRegio έχει καταστεί πιο δεκτική και πιο εντατική. Γίνονται πιο πολλές συναντήσεις σε επίπεδο γενικών διευθυντών. Έχουμε καταλόγους, checklists που χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προετοιμάζονται με την υποστήριξη της DigiCompt και τις οποίες ε, χορηγούμε και στους εθνικούς ελεγκτές. Όπως σας είπαμε ήδη, η Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ είναι μια διεύθυνση στην οποία συμβουλεύεται πολλοί κόσμος για το κατά πόσον υπάρχει συμβατότητα των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε περίπτωση μεγάλων έργων. Προσπαθούμε δε να συντονιστούμε όσο πιο πολύ να συντονίσουμε μάλλον την εποπτεία των μεγάλων αυτών προγραμμάτων μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης ΚΟΜΠ και των συναδέλφων μας στην Γενική Διεύθυνση Ρίτσιο, παρά το γεγονός ότι η οι διαδικασίες αμφότερες έχουν διαφορετικούς στόχους. Οι τελευταίες αιτήσεις εκθέσεις που μας έδωσαν οι Εθνικές Αρχές το Φεβρουάριο σε ό,τι αφορά τις ε, δαπάνες μεταξύ του Ιουλίου 2016 και τέλη Ιουνίου 2017 αναφέρουν 35 σφάλματα σε ό,τι αφορά την κρατική ενέσχυση που σχετίζονται με την έλλειψη ή το μη σεβασμό των διδάξεων για την εποπτεία, μη κοινοποιούμενη κρατική ενίσχυση ή ε, λανθασμένη εφαρμογή των προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης και επίσης η λανθασμενη εφαρμογη των προγραμματων ε, κρατικης ενισχυση και επισης η υπερβαση των οριων de Να κλείσω λέγοντας το εξής. η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και οι κρατικές ενισχύσεις όχι μόνο είναι συμβατέ, αλλά συνδέονται και στενά. Και για την περίοδο μετά το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται ακόμα πιο πολύ σε μέτρα για την προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε λιγότερο Αναπτυγμένε περιοχέ, Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξει η μεγαλύτερη επικέντρωση στα μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και πρωτοβουλίε Αυτό Ενδεχομένω να αυξήσει και τι κρατικέ ενισχύσει, Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περίπλοκοι οι κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει για τι ε, αρχέ και ότι υπάρχουν πολλοί έλεγχοι από τι εθνικέ αρχέ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ελεκτικό Συνέδριο και ότι οι διαδικασίε μπορεί να μην είναι οι ίδιες μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης ε, Κομ και Ρέτζιο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι αλληλοσυμπληρούμενε, αλληλοσυμπληρωματικές. Θα συνεχίσει, λοιπόν, η συνεργασία μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο τέταρτο και τελευταίο μιλητή μα τον κύριο Ρόιτερς, για τις ε, μεταφορές στη ΓΑΜΑ ΜΟΥ, για ε, μεταφορές ευφυής κτλ. Αγαπητέ Πρόεδρε, και κύριοι αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα. Θα μπορούσα να μην πω πολλά από αυτά που έχω προγραμματίσει να πω γιατί τρεις προλαλήσαντες με κάλυψαν. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΦ και τις επενδύσεις στα διεθνή διευρωπαϊκά δίκτυα, είναι σημαντικές οι επενδύσεις βλέπετε τα ποσά και σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλες επενδύσεις, ιδίως τώρα που μιλάμε για τη μετάβαση στην ευφύ κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Κάτι σημαντικό ιδίως για τις αστικές περιοχές. Συστημική είναι η στοχεία της αγοράς ε, στον τομέα των μεταφορών και έχουμε και υψηλό επιθετικών ε, εξωτερικών στοιχείων ε, χωρίς αυτό αυτή τη δημόσια παρέμβαση δεν θα μπορούσε η πολιτική για τα ευρωπαϊκά δίκτυα να πετύχει. Έχουμε τώρα τον κανόνα ε, ΣΕΦ, τον κανονισμό ΣΕΦ που ορίζει τους κανόνες για τη χρηματοοικονομική υποστήριξη σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Μόνο υποστήριξη υποδομών παρέχει το ΣΕΦ, 70% για το σιδηρόδρομο. Δεν είναι κρατική βοήθεια, αλλά ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται απευθείας η Κομισιόν. Το είπε και ο Κόπμαν η υποστήριξη γραμματοδότηση από τα κράτη-μέλη μπορεί να έχει να κάνει με κρατική βοήθεια, αλλά οι συνδρομικέ υποδομέ, για παράδειγμα, που χρηματοδοτούνται κατά κόρον από αυτό το μέσο, δεν καλύπτονται. Ξεκάθαρα λοιπόν τα είπαν οι προλαλήσαντες ε, για το ΣΕΦ. Όμως, Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Στο πλαίσιο του ΣΕΦ πάντα. Τα χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχει σημαντική αύξηση της χρήσης των μέσων αυτών για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα βασίζονται πάντοτε σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση για να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και για να υπάρχει συμβατότητα με του κανόνε περικρατικών ενισχύσεων. Συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου μα από την Γαμαλτά Μπάτ και ΕΚΦΙ για το InvestEU Program. Ένα πρόγραμμα που το ανέφεραν προλαλήσα Και έτσι μπορώ να καταλήξω σε αυτή την πολύ σύντομη παρέμβασή μου. ότι τηρούμε όλη σχετική νομοθεσία και θέλουμε να υπάρχει συνεκτικότητα με τη, και με το δανειακό μέσο ε, και με τις κρατικές, ε, τις κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Ελπίζω να καταλάβατε και να έχετε έτσι μια πιο πλήρη εικόνα για το τι ισχύει ε, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Πάρα σε ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα Ο εισηγητής. Ε, Η εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους ομιλητές που μας έδωσαν κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προσεχή πολίτη ε, προπολογισμού. Σίγουρα η συζήτηση στο μέλλον θα είναι πιο ζωντανή γιατί θα έχουμε μείωση σε σημαντικές πολιτικές. Επίσης θα έχουμε νέες πολιτικές. Και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και πώς θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ερώτησή μου κυρίως είναι η εξής. έχουμε αυτό το Invest ε, in You, θα πρέπει να λάβει πώς τα διάφορα αιτήματα και άλλους ε, ίσως χρηματικοπούς ε, διαμεσολαβητές. Το είπε και η κυρία από τη Γαμαδελτα Ρέγγιο. έχουμε τον νέο προπολογισμό. Πώς θα προχωρήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θα διαμορφώσουν τις ενισχύσεις και τη βοήθεια θα παρέχει ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό στα διάφορα αυτά έργα. Πώς θα καθορίσουμε για να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, εγκαίρες κτλ. ή αν δούμε βελτιώσεις να τις προβάλλουμε eh, digamos, vía un, un compromiso mayor. να μην έχουμε προβλήματα. Πώς λοιπόν από το Κοινοβούλιο μπορούμε να βοηθήσουμε. Να προωθηθεί το όραμα αυτό και να μην υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα. Κάθε φορά που έχουμε νέε δεσμεύσει στα κράτη-μέλη, Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με κάποιους κανόνε εξαίρεση από τους κανόνες ε, κρατικών ισχύσεων κτλ. Δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια. και υπάρχουν ε, ανώμαλες καταστάσεις και μέσα και έξω. Όχι γιατί δεν εφαρμόζονται οι κανόνες, αλλά γιατί δεν δίνεται σωστή ενημέρωση στους πολίτες. Και είμαστε και στην τελική ευθεία πριν τις ευρωεκλογέ. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πρέπει να είναι πιο διαφανής η εφαρμογή των κανόνων αυτών. και των επιπτώσεων που έχουν. ώστε η πληροφόρηση να είναι σαφής. Για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προπολογισμού πρέπει να υπάρχει διαφανής πληροφόρηση. Και αυτό είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν και άλλα. Σε ό,τι αφορά όλα τα μέτρα, τα οικονομικά που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και τα βλέπουμε όλα αυτά, εκεί δεν έχουμε την επαρκή πληροφόρηση. ή να πω την ξεκάθαρη πληροφόρηση για να υπάρχει διαφάνεια. Όχι από πλευρά κομισιό, από αλλά μιλάω για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τα σχετικά. Por, por las exenciones de bloque. θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους νέους αυτούς κανόνες. και πώς επηρεάζεται η οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η χρηματοδότηση γενικώ. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και για έργα πάρα πολύ σημαντικά που συνιστούν στην αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Χρηματοδοτείται από όλου, αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν ποιο χρηματοδοτεί τι και πότε. Okay, I think the main question there was... Uh, Βασικό ερώτημα, νομίζω και ζήτημα, είναι πώς θα είναι πιο ξεκάθαρη και διαφανείς οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος, κύριε Κούπμαν. Thank you uh, very much for that. Uh, ναι, ευχαριστώ. Ήταν πολύ εύστοχο το ερώτημα. Τρει απαντήσει. Ή μάλλον τρία σκέλη θα μπορούσε να έχει απαντησή Σε ό,τι αφορά το MSTU, καταρχάς, το κ. Βάλμπρουκ. Τι θα κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα. Τις κανόνες κρατικών ενισχύσεων θα τους θέσω πολύ ξεκάθαρα και θα τους συμπεριλάβουμε ε, στους κανόνες ε, της επενδύσεις. Ώστε να υπάρχει αυτόματα συμφωνία. Αυτό θα είναι μεγάλη απλούστευση. Κανόνας κρατικών ενισχύσεων, όπως και κανόνας του UNVEST θα είναι δημόσια γνωστή και διαθέσιμη. Η ΓΑΜΑ ανταγωνισμό θα το κάνει αυτό στον κανονισμό περί γενικού μπλοκ ε, εξαιρέσεων, θα επικαιροποιηθεί και όλοι οι πολίτες και επιχειρήσεις των κρατών μελών θα μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση σε αυτό το rule book. Άρα θα είναι ξεκάθαροι κανόνες. Ένα άλλο ερώτημα που θέσατε ήταν Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τελικά τι δαπανούν τα κράτη-μέλη. Γιατί μιλάμε για ένα ε, μιλάμε για μια εξαίρεση. Αλλά παρόλα αυτά, παρότι θα έρθουν στι Βρυξέλλες, θα πρέπει κάπως να τα εξηγήσουν. Στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού που ανέφερα, το καλό είναι ότι είναι υποχρεωτικό πλέον κάθε μεμονωμένο μέτρο κατοικών ενισχύσεων πάνω από 500.000 ευρώ θα πρέπει να δημοσιοποιείται σε ένα μητρό διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΑΜΑΤΑΚΟΜ διαχειρίζεται το σχετικό αυτό μητρό και έχουμε πάνω από 40.000 λίματα ήδη. Βλέπετε, βλέπετε ποιο είναι ο δικαιούχο, το ποσό τη ενίσχυση ε, για το σκοπό που δόθηκε. Άρα υπάρχει διαφάνεια για όλου. Και θα έλεγα ότι και γι' αυτό στο Κοινοβούλιο πληροφορίε που είναι σημαντικέ. Και περιμένουμε όσο προχωρούμε να βελτιώνεται στο πλαίσιο της νέας περίοδου προγραμματισμού αυτή η ενημέρωση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση από πλευράς μου που συνδέεται Νομίζω η κυρία Φερνάντες Γιούτς μας έδωσε ένα κατάλογο των σφαλμάτων και τους λόγους στους οποίους οφείλονται. Ένας από ένα από τα σφάλματα ήταν ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Γνωρίζετε γιατί τα κράτη-μέλη δεν κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι αυτό ή θελημένο που φυσικά είναι λάθος ή δεν γνώριζαν τους κανόνες. Και αν όντως περί αυτού πρόκειται, φυσικά θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στην επικοινωνία. Για ποιο λόγο δεν κοινοποίησαν την κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν κοινοποιήθηκαν ε, οι πληροφορίες ε, αρκετά νωρίς. Ε, όμως ε, διαπιστώσαμε ότι στο παρελθόν δεν ήταν θελημένο, ήταν λάθος ερμηνεία των κανόνων. Κάποιες φορές ο δικαιούχος δεν είχε καν καταλάβει πως ήταν κρατική ενίσχυση ή μπορεί να πιστεύουν ότι είναι εξαιρε... εξαιρούμενοι, ενώ δεν είναι. Αλλά δεν έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες. Δεν έχουμε ποτέ πάντως συναντήσει η θελημένη μη κοινοποίηση. Ωραία, σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανείς άλλος να ζητά το λόγο, οπότε θα κλείσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και που ε, απαντήσατε στις ερωτήσεις. Ήταν μια καλή αρχή σε αυτή τη μας την ακρόαση και σας ευχαριστώ και πάλι από πλευρά της Επιτροπής μας. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη συζήτηση όπου ο τίτλος είναι «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν τους κανόνες». Και εδώ έχουμε τρεις συναδέλφους που θα κάνουν εισηγήσει. Τα ονόματα των προηγούμενων ομιλητών ήταν σχετικά απλά, αλλά τώρα δυσκολεύομαι πολύ περισσότερο. Πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Έστερ Σούλτ, που είναι, είναι αναπληρώτρια επικεφαλής του τμήματο τη ε, της ε, αρχή αρχής EFDR της Βάδης Βουτεμβέργης. Παρακαλώ λοιπόν έχετε το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Εισηγητρία, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, κύριε και κύριοι. Να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ σε αυτή την ακρόαση και χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνω το λόγο για να μπορέσω να μιλήσω και από πλευρά τη Βάδα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ε, κάποια άλλη μικρά στατιστικά στοιχεία, αν μου επιτρέπετε. Βλέπετε το μερίδιο των κρατικών ενισχύσεων για το 2016 σε ό,τι αφορά το σύνολο. Μιλάμε σε επίπεδο 8% στο ευρωπαϊκό επίπεδο, 4% σε επίπεδο των συνολικών ταμείων και ενισχύσεων στη Γερμανία. Θα δούμε λοιπόν, πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, είναι όντω πρόκειται για περικρατική ενίσχυση ή όχι. τις ε, δυσκολίες που βλέπουμε στα πλαίσια της ενίσχυσης EFRE. E. Καταρχάς έχουμε τις ε, πρωτοβουλίες και όλα τα επίπεδα πρωτοβουλίας με τη δημιουργία ε, γνώσης, μεταφορά τεχνολογίας μέχρι και εταιρείε τεχνολογίας ε, και μετά σε δεύτερο επίπεδο, σε επίπεδο δήμων και επιχειρήσεων. Και από αυτούς τους δύο τομείς, λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω στοιχεία. Μία μικρή επισκόπηση. Ο τοπικός χαρακτήρας των επενδύσεων, καταρχάς ε, ύστερα τομείς ενίσχυσης με δύσκολο έλεγχο ενίσχυσεων, για παράδειγμα, υποδομές, ε, δομές υποστήριξης για επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες ενέργειας και ένας γενικότερος ε, τομέας η άμεση και καταναμημένη παροχή μέσων, τα κριτήρια τα που εφαρμόζονται για το κατά πόσο πρόκειται για ενίσχυση. Τα γνωρίζετε. Μια επιχείρηση θα πρέπει να ζητάει να χρησιμοποιούνται κρατικά δημόσιοι πόροι, να υπάρχει προνόμιο, να υπάρχει επιλεκτικότητα, επιλεξιμότητα και τέλος να μιλάμε και για υπονόμευση του ανταγωνισμού στα πλαίσια του κράτους μέλους. Το τελευταίο κριτήριο μας οδηγεί και στο θέμα του τοπικού χαρακτήρα της εφαρμογής των επενδύσεων. Εδώ λοιπόν αναρωτιόμαστε κατά πόσον οι υπηρεσίε και τα προϊόντα παρέχονται σε ένα περιορισμένο χωρικά, σε ένα περιορισμένο χωρικό, κατά πόσον υπάρχουν πελάτες από άλλα κράτη-μέλη και κατά πόσον υπάρχουν διασυνοριακές επενδύσεις. Και ο έλεγχος ε, αυτού του κριτηρίου λοιπόν καθαρίζεται από τον τοπικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι δύσκολος να οριστεί Υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου διαπίστωσε για παράδειγμα ότι λόγω του τοπικού χαρακτήρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για στρέπλωση του εμπορίου και του ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά για μας θα ήταν ευκταίο να υπάρχει συστηματική παροχή των στοιχείων αυτών. Για παράδειγμα στην κοινοποίηση της ενίσχυση. Ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά τις υποδομές για επενδύσεις. Ε, υπάρχουν τρία επίπεδα τα οποία εξετάζονται στις ενισχύσεις ε, φορέας, ε, πάροχος και χρήστης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτή η επένδυση, αυτός ο πόρος μπορεί να περάσει από τον φορέα μέχρι τον χρήστη. σε επίπεδο χρήστη, είναι δύσκολο να εστιαστεί το στοιχείο της ενίσχυσης και να καθοριστεί όταν παρέχεται μία σειρά υπηρεσιών, για παράδειγμα, τα οποία σωρευτικά δεν μπορούν να καθοριστούν και δεν γνωρίζουμε τελικά πόσα θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια ύπαρξης της ε, υποδομής. Θέλουμε λοιπόν ε, σε επίπεδο χρήστη να υπάρχουν πιο πολύ εφαρμόσιμε πρακτικές. Και σας δείχνω την ίδια εικόνα λοιπόν άλλη μια φορά. Εδώ κοιτάμε πιο πολύ τον φορέα και τον ε, διαχειριστή. Εδώ είναι ιδιωτικά άτομα, είναι Ενδεχομένω να προκύψουν σφάλματα στην εφαρμογή του σχετικής νομοθεσίας και Υπάρχει το ερώτημα του κατά πόσον συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς και κατά πόσον είναι σωστή τελικά η τιμή. Και εδώ έχουμε και άλλη πτυχή σε ό,τι αφορά την κοινιοποίηση. Αλλά και το ορόσημο βάσει μέσης τιμής είναι μια πρακτική η οποία ούτε ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και δύσκολη στην εφαρμογή της ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή, την υπολογισμό της, ε, της τιμής της αγοράς. Παρόμοια προβλήματα έχουμε και για τις υποδομές ενίσχυσης ε, επιχειρήσεων, Μικρομεσές επιχειρήσεις για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την παροχή υποστήριξης για την καινοτομία, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε κατά πόσον αυτές οι δομές ε, είναι ελεύθερες από ενισχύσεις ε, και επίσης είναι δύσκολο να καθορίσουμε κατά πόσον οι επιχειρήσει ε, χρησιμοποίησαν πραγματικά ενισχύσεις και εδώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέχονται εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις μια άλλη πτυχή ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε ενέργειε και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Συχνά υπάρχει προσαρμογή στην αρχή τη προστιθέμενη κόστους. σε σχέση δηλαδή με τις ε, παραδοσιακές ε, επενδύσεις υπολογίζονται το επιπλέον κόστος το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της άμεσης ενίσχυσης. Είναι λίγο περίπλακο το σύστημα και εδώ θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει απλοποίηση για να υπολογίζεται το ποσοστό στο οποίο αναλογεί κάτι και ενίσχυση. Αν είναι τελευταίο θέμα. Σε ό,τι αφορά την ε, άμεση και διερεμένη διαχείριση μέσων και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις. Θέλουμε συγκρίσιμα project και έργα. Θα πρέπει να είναι ίση η αντιμετώπιση των προγραμμάτων τα οποία περνάνε από κοινή διαχείριση ή τα οποία είναι στην πολιτική διαχείριση των κρατών μελών. Ένα παράδειγμα, η σφραγίδα αριστείας. Το ακούσαμε σε διάφορες περιστάσεις από διάφορους ομιλητές. Το πρόβλημα που είναι ότι στην αποκλειστικη διαχειριση των κρατων μελων ενα παραδειγμα η σφραγιδα αριστειας το ακουσαμε σε διαφορες περιστασεις απο διαφορους ομιλητες το προβλημα που ειναι οτι στην οριζοντα 2020 παρέχονται και μπορούν να παρέχονται καλύτεροι όροι σε ό,τι αφορά τις ε, άλλες διατάξεις όπως η EFRE, η οι διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται μια καλή λύση προκειμένου να υπάρχει αναρμόνιση των εργαλείων σε ό,τι αφορά της, ε, την ε, άμεση και διαιρεμένη διαχείριση και χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους όρους ε, για τις άμεσες ενισχύσεις και σε αυτά θα ήθελα να περιοριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας. Κυρία Γεωργοπούλου τώρα, για πιστικέ υπηρεσίε για κρατικέ ενισχύσει Υπουργείου Οικονομικού ε, στην Ελλάδα. Έχετε το λόγο κύριε Γεωργοπούλου. Dear Mr. President, dear Mrs. Rapporteur, dear colleagues, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί αγαπητές ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε την συνοχή και τον ανταγωνισμό από διάφορες απόψεις. Ε, προσπαθεί η αρχή μας να ευθυγραμμίσει τα... Ε, τις προσπάθειες εδώ. Θα εστιαστώ λοιπόν στις διάφορες μεθόδους, στους διάφορους κανόνες, στις διάφορες πολιτικές και τις διάφορες διαδικασίες των ε, δύο γενικών διευθύνσεων. Η μέθοδοι. Πώς ε, υπολογίζουμε δηλαδή τα ποσά στήριξης για τα διάφορα project. Προβλέπουμε τον υπολογισμό ε, με συγκεκριμένες μεθόδους που είναι όμως απαραίτητα κοινέ για να μπορέσουμε ε, να συνοηθούμε μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Επί, επί την, επιπλέον, όταν έχουμε δύο project με το ένα μεγατική ενίσχυση, το άλλο όχι, ε, το κάνουμε αυτό με συγκεκριμένη ε, προσπάθεια. For project generating profits, with a total Αυτό όταν είμαστε κάτω από τα 1 εκατομμύριο το προσπαθούμε αυτό. Όταν όμως ε, ε, υπάρχει διπλή χρηματοδότηση τότε είναι πολύ πιο περίπλοκο. Δυστυχώς η ομιλήτρια μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε να την ε, παρακολουθήσουμε. Ε, διαβάζει το κείμενό της και είναι σχεδόν αδύνατον για τους ερμηνείς να παρακολουθήσουν. private contribution, which is state funding, would also be considered as state aid. So, in this case, the state... Λοιπόν, ε, το κράτος προσπαθεί να πάρει μια συμβολή μέσω ενός δανείου, ακόμα και αν αυτό δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά διαφορετικούς κανόνες, ε, το CPR ξεκίνησε και έθεσε την ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών τον Ιούνιο. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη πριν να υποβληθεί η αίτηση. Σύμφωνα με τους κανόνες ε, περί κρατικών ε, ενισχύσεων, είναι επιλέξιμο αυτό πριν την αίτηση. Εάν όμως ε, ε, έχουν γίνει ήδη δαπάνες, τότε το project δεν είναι επιλέξιμο για ενίσχυση. Αυτό συχνά αποτελεί ένα ε, πλεονέκτημα και ένα κίνητρο. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε για την ε, περίοδο επιλογής μέχρι το τέλος ε, του 2023, του κανονισμού δηλαδή ΕΣΥΦ, ώστε να αποφύγουμε τα ήδη κοινοποιημένα project τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του ε, ΕΣΥΦ. Σύμφωνα με τους κανόνες περικατικών ε, ενισχύσεων, οι ε, οικονομικοί ε, διαμεσολαβητές θα πρέπει να επιλέγονται μέσω ενός καθαρού διαγωνισμού. Δεν έχουμε ανοιχτό διαγωνισμό ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα ότι η εφαρμογή ενός ε, βραβείου εντός ε, θα εξαλείψει την, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ενισχύσεις. Για τις υποδομές υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δύο μονάδες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής ε, μιας υποδομής. Διαφορετικές δυνατότητες επιλογής. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα project τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στα εγκεκριμένα ε, επιχειρησιακά προγράμματα, λειτουργικά προγράμματα, δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό αίτημα και αυτό αυξάνει το, τελικό, το διοικητικό άχθος νομοθετικής απαιτήσεις. Το διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδοτούν ε, τις περιοχές που ε, συναντούν δυσκολίες. Η ομιλήτρια συνεχίζει να διαβάζει το κείμενό της πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να την παρακολουθήσουμε δυστυχώς. Οι κανόνες περικατικών ενισχύσεων επιβάλλουν μία επιλεκτική προσέγγιση και αυτό έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή της στρατηγικής. Διευκρινίζονται τομείς και, περιφέρειες όπου χρειάζεται συγκεκριμένη ανάπτυξη. Ας πούμε, κατάρτιση για τους ε, υπαλλήλους μπορεί να θεωρηθεί κατοική ενίσχυση προς εταιρείε που τους απασχολούν, ακόμα και αν οι εργαζόμενοι αυτοί δουλεύουν σε τελείως διαφορετικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, διαφορετικού είδους κρατικές ενισχύσεις μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή, γιατί δεν είναι τόσο ελκυστικές για τις επιχειρήσεις. Οι δύο πολιτικές είναι κάπως διαφορετικές. Από τη μία πλευρά έχουμε την πολιτική συνοχή που στόχο έχει να αναπτύξει την ε, ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως οι δραστηριότητες καινοτομία πιο κοντά στην αγορά στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Regarding procedures, a very important problem is the need to deliver a lot of information to the EU for both Δίνονται πολλές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Οι εθνικές αρχές πρέπει να συμπληρώσουν διάφορες, ε, διάφορα έντυπα Προτείνουμε την ενοποίηση αυτών των ε, μέσων, προωθώντας την ε, διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Of just one approval decision which cover both... Δυστυχώς, όπως σας είπαμε, ήδη η ομιλήτρια διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε. Monitoring checks are carried out by different authorities on the same issues. We propose to mainstream at least all the evaluations. Προτείνουμε την ευθυγράμμιση των ε, διαδικασιών αξιολόγησης δημοσιότητα και διαφάνεια. Αυτά πρέπει να προωθηθούν και πρέπει να συντονιστεί αυτό ανάμεσα στα ιδιωτικά ταμεία και τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό είναι προφανές. The DG Agri approach. Milestones and procedures. OP sets indicators, milestones, which are important to achieve since they are related to payments performance reserve allocation and other important issues. However, for measures which require notification, DGCOM, to DGCOM, procedures of the takes off. Η διαδικασία αυτή συχνά παίρνει έξι και περισσότερους μήνες. Και δεν επιτυχάνεται τίποτα λόγω της ε, καθυστέρησης που υπάρχει στη διαδικασία ανταγωνισμού. χρειάζεται περισσότερη ε, ε, απλοποίηση, ας πούμε απλοποιημένα σε επιλογές κόστους. Μέχρι την έγκριση της τροπολογίας Δίμπερ δεν υπήρχε νομική βεβαιότητα όταν χορηγείται η ενίσχυση και γινόταν υπο, τον υπολογισμό μιας απλοποιημένης διαδικασίας. Η DG Regio και η DG Employment θα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν αυτήν την απλοποιημένη επιλογή κόστους ε, όταν αξιολογούμε την ενίσχυση στην καινοτομία για τις τοπικές υποδομές, όταν είναι πραγματικά τοπική κόσμο χαρακτήρες και αποκλείεται η κρατική ενίσχυση, αν πρόκειται για μία τοπική υποδομή ε, που καλύπτεται από το 56 της Τζίμπετ. Αν και τέτοια προγράμματα σχετίζονται με την κρατική ενίσχυση, πώς να αξιολογείτε τελικά. Στη local. Last but not least are the ETC projects. ETC projects require cross-border cooperation and partners from different countries. Η ομιλήτρια δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Μιλάει, γρα, διαβάζει ένα γραπτό κείμενο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. In the view of the low budget and the objective of these projects, we propose to examine the possibility to extend future, to exempt future ETC type actions from state aid rules at least to some extent. As in conclusion, we have to say that although many steps have been taken, Πολλά βήματα έχουν γίνει. Πολλά όμως πρέπει ακόμη να γίνουν. για να υπάρχει αναρμόνιση. Wow. Uh, we wanted to talk about uh, difficulties faced by member states. Ακούσαμε μια πολύ μακρή κατάλογο των δυσκολιών που έχουν αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Ίσως στο τέλος του μάτους. Κάποια από αυτά τα θέματα να τύχουν μια απάντηση, ξέρω αν κάποιο συνάδελφο. Και ο Σκούπμαν ίσως. Τρίτη παρέμβαση. Πάμερα Ρόμπελ. Από το Υπουργείο Παρακολούθηση Κατοική Βοήθεια στην Πολωνία. Uh, uh, Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ και που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω για τα κονδύλια εύση. Πολύ σύντομη θα είναι η παρουσίασή μου. Ουσιαστικά υποχρεωμένη να συμφωνήσω με όλα όσα είπαν η Γερμανίδα και η Ελληνίδα συνάδελφος. Το ευχαρι... Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μου κάνετε πιο εύκολη τη δουλειά μου. Παρ' όλα αυτά θα σας ε, μεταφέρω την πολωνική εμπειρία. Οι συνάδελφοί μου λοιπόν μάλλον η κυρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εστίαση στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο το παρελθόν, που είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για το σχεδιασμό του μέλλοντος, να αποφύγουμε δηλαδή τα λάθη του παρελθόντος. Κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικαίου περιανταγωνισμού και τα ταμεία του ΕΦ ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής είναι δύο δέσμες ε, κανόνων δύο ευρωπαϊκές πολιτικές και δύο διαφορετικές απόψεις. Η πρόσφατη τάση είναι οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων να θεωρηθούν εμπόδιο σε ό,τι αφορά ε, τη διάθεση των κονδύλων ε, συνοχής. Η εφαρμογή μια ε, πολιτική δηλαδή απειλεί την εφαρμογή μια άλλη πολιτική, αντίστοιχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό είναι επικίνδυνο επειδή συμμετείχα ε, στα τεκτενόμενα για τις κρατικές ενισχύσεις, ε, νομίζω ότι αυτή η προοπτική ε, μου έρχεται λίγο κάπως πιο φυσικά. Γι' αυτό θέλω να προσθέσω ένα άλλο ζήτημα, ένα άλλο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ταμείων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, πόση κρατική βοήθεια παρέχεται την Ένωση και τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό στο δοκινοτικό εμπόριο και στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. κ. Κόπμαν, και τον ευχαριστώ για αυτό, μίλησε για το ποσοστό των σχεδίων και έργων που υπάρχει συνδύση τόσο κρατικών ισχύσεων είναι από 20 30%. 20 μάλλον με 25%. 27% των δαπάνων στην Πολωνία και 22% όλων των έργων έύση καλυπτώνται από το τομέα αυτό των κρατικών νησιών, αλλά δεν είμαστε ίσως το καλύτερο παράδειγμα. Περιορισμένος ο χρόνος. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τα βασικά προβλήματα που είχαμε σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση προς κανόνες ε, σε τα ταμεία, τα κονδύλια του Ταμείου ΕΦΣΥ. έχω κάνει αυτή τη διάκριση στις κατηγορίες αυτές που είπα. Δύο είδη κανόν, διαφορετικοί στόχοι, διπλές υποχρεώσεις. Όλα αυτά έχουν ε, και κάποιες επιπτώσεις. Το ότι έχουμε δύο δέσμες κανόνων, για παράδειγμα, δεν σημαίνει πάντα βέβαια ότι είναι αντιφατική μεταξύ τους. Όμως το ότι έχουμε δύο ορισμούς για την ίδια είναι για παράδειγμα. Καινοτομία, ένα έργο, ένας δικαιούχος δεν είναι συγκλίνων κατάλογο σε αυτό το επιλέξιμο κόστος. Η σχολεία στην εφαρμογή. Δύο διαφορετικοί στόχοι. Γιατί έχουμε την πολιτική συνοχή αφενό και την πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Στόχο πολιτική ανταγωνισμού ποιο είναι, να προστατεύσει την εσωτερική αγορά και να εξασφαλίσει του ίδιου όρου και συνθήκε για όλους τους ε, φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Στόχος της πολιτικής συνοχή είναι οι ίδιε συνθήκες και οι ίδιοι όροι, αλλά να εξισωθούν αυτοί. Άρα είναι αναγκαίο να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η εξίσωση των όρων, χωρίς όμως να έχουμε υπερβολικά ευνοϊκή μεταχείριση κάποιων φορέων από, λιγότερες, αναπτυγμένε Τρίτη κατηγορία οι διπλές υποχρεώσεις και καθήκοντα. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε διοικητικό άχθος, Περιβολικό σε πολλές περιπτώσεις, που στα άκρα θα μπορούσε να οδηγήσει και στην παρέτηση από ένα αναπτυξιακό έργο. DG Comp, DG Regio ε, δικαιολογούν ε, τις διαδικασίες τους. Προφανές αυτό. Το θέμα είναι όμως, μπορεί να γίνει κάτι για να υπάρχει εναρμόνιση αυτών των διαδικασιών. Τώρα θα ήθελα εν συντομία να σας δείξω ακριβώς κάποια παραδείγματα για να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, και όχι μόνο στην Πολωνία, το ανέφερε η Γερμανίδα συνάδελφος, είναι η διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων ε, έργων λόγω της πηγής χρηματοδότησης. Έχουμε κάποια πράγματα με κεντρική διαχείριση και κάποια άλλα ε, κονδύλια που είναι στη θέση των κρατών μελών. Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και στην άλλη έχουμε έργα τα οποία είναι εκτός ε, πεδίου εφαρμογή. Άρα οι δικαιούχοι προτιμούν την κεντρική διαχείριση γιατί η χρηματοδότηση δεν εμπίπτει στο επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων. Όπως μπορείτε λοιπόν να δείτε μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για ένα είδος αντιπαλότητας μεταξύ προγραμμάτων. Επίσης, δεν είναι συνεκτικοί οι ορισμοί, ε, τα επιλέξιμα στα πάνες, καινοτομία κτλ. Άρα δεν είναι σαφείς οι κανόνες και δεν υπάρχει και ασφάλεια δικαίου λόγω αυτού. Επίσης, η μέθοδος του απιστευμένου κόστος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται όπως είπε Ένα άλλο θέμα είναι μια διαφοροποίηση, ένα κενό ε, που έχουμε σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και η ένταση της βοήθειας ε, στα project που χρηματοδοτούνται ε, σε κρατικό επίπεδο. Δεν θα επισέλθω σε τα είπε η Ελληνίδα συνάδελφος. Already mentioned briefly the gap between... Μίλησε για ένα χάσμα μεταξύ πολιτική συνοχή και πολιτική ανταγωνισμού. Θα ήθελα να σα δείξω αυτό το χάσμα στην πράξη ε, πώ έχει και τι επιπτώσει μπορεί να προκαλέσει. Για την Πολωνία πάντα. Δύο καταστάσεις. Θα σας περιγράψω. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα πρώτα. Έχουμε κάποιε δραστηριότητε που τις εγκρίνει η ΓΑΜΑ η Κομισιόν, στα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί όμω αυτέ τι δραστηριότητε αν δεν είχαμε το πρόβλημα με τα κριτήρια επιλεξιμότητα. Κανόνε κρατική βοήθεια δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση στην Κομισιόν. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Ακόμα στη διαδικασία της υποβολή των προγραμμάτων. Αυτό αφορά τα συστήματα θέρμανσης ψήξης που δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά. Δεύτερο παράδειγμα για την περίοδο προγραμματισμού 7-14. Όταν είχαμε την αλλαγή των κανόνων περί κρατικής βοήθειας και ο τομέας ενέργειας εξαιρέθηκε από τις περιφερειακές ενισχύσεις, στη φάση ε, κατάρτισης ε, του επιχειρησιακού προγράμματος έγινε αυτή η αλλαγή στη μέση της ε, εφαρμογής δηλαδή της εκτέλεσης και αυτό βέβαια δημιούργησε προβλήματα. Υπάρχουν κάποια έργα που χρηματοδοτήθηκαν στην αρχή της περίοδου αυτής προγραμματισμού και άλλα τα οποία είχαν εφαρμοστεί με το προηγούμενο καθεστώς και άλλα που ήταν στο τελικό, στην τελική φάση και έπρεπε να αντιμετωπιστούν τελείως διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το επιλέξιμο κόστος και την ένταση βοήθειας ή ενίσχυση. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. μήνες και χρόνια καθυστέρησης. ούτε την ανάγκη να υπάρχουν εξατομικευμένε διαδικασίε να αφισβητούμε, ούτε ε, το κατά πόσο είναι θεμητό ή όχι να γίνεται κάτι τέτοιο. Και σίγουρα χρειάζονται έλεγχοι, παρακολούθηση, ιδίω έχοντα υπόψη ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερη εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, λόγω του κανονισμού για τα block exemptions. Όμως, καλό θα ήταν να υπάρξει κάποια αναρμόνιση. Πρέπει μια μορφή κοινοποίηση μπορεί να πληρεί τα κριτήρια και των δύο γενικών διευθύνσεων. Και έτσι να μην χρειάζονται δύο. Για να συνοψίσω και να σας πω τι αποτέλεσμα έχουν όλα αυτά για την Πολωνία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει εναρμόνιση και καλύτερο συντονισμό. Και επαναλαμβάνω αυτά που είπαν ε, οι προέλισσα συναδελφοί μου. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε κανόνες και διαδικασίες που είναι αιτιολογημένες, αλλά ο στόχος είναι να επανεξετάσουμε και να προβούμε σε τυποποίησεις όπου αυτό είναι δυνατόν. Κάποιες παρατηρήσεις λοιπόν τώρα από τα πολυελληνικά αυτά παραδείγματα, σύντομα. Πρώτη, παρατήρηση. είναι να υπάρχει μια εναρμόνιση ε, τη διάρκεια κανόνων κρατική με τι περιόδου προγραμματισμού για το ΕΣΥΦ και την αρχή ε, του ΝΙΣΥΝ. Επίσης, για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θέλουμε να γίνεται μια αρχική επαλήθευση ό,τι αφορά την κρατική βοήθεια. Ένα fast track, μια ταχεία διαδικασία, παραδείγματο χάρη για την ερμηνεία των κανόνων αυτών για τα προγράμματα ESIF ή η αμοιβαία αναγνώριση αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων των ελέγχων ή αναθεώρηση και ενοποίηση των ορισμών. Και αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Ορισμένες από αυτές τις παρατηρήσεις, οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα σημαίνει ότι ήταν καλές ιδέες αυτές. Αυτά, ευχαριστώ. Thank you. Another, uh... Σας ευχαριστώ και άλλη μία εξαιρετική παρέμβαση με πολύ καλά παραδείγματα. Είπαστε στην αρχή ότι θα είστε σύντομοι, αλλά μιλήσατε παραπάνω από ότι τη για άλλε συναδελφοί, αλλά δεν πειράζει γιατί είχαμε λίγο χρόνο και έχουμε λοιπόν πολλά παραδείγματα από δυσκολίε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κούπμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε κάποια από τα θέματα αυτά, τα οποία είναι πολύ περίπλοκα και κάποια θέματα που μπορούσατε να μας δείξετε σε ό,τι αφορά κάποιες διευκρινήσεις ε, για το ποιο δικαιούται και τι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από τα κρατημέλη που έκαναν λεπτομερείς παρουσιάσεις. Προφανώς δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομερείς για κάθε θέμα που θίξατε και δεν νομίζω ότι άλλωστε θα είχε νόημα γιατί όπως είπαν και οι συνάδελφοι δικαίω σε κάποιες περιπτώσεις τα θέματα αυτά είναι θέματα του παρελθόντος, όχι τόσο πολύ του μέλλοντος. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εξηγήσουμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα θέματα θα τα επιλύσει το νέο που το Το ε, δεύτερο θέμα, ένα βασικό σημείο ότι οι δύο πολιτικές έχουν σχετικά διαφορετικούς στόχους και η διαπαφή μεταξύ των πολιτικών είναι μάλλον μικρή. Στην Πολωνία ίσως να είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι το Μεσόωρο. Αλλά όπως μας είπε η συνάδελφος από τη Βάδη Δεμέργη, εκεί η αλληλεπικάλυψη είναι 4%, στην Πολωνία ίσως είναι 20%, κατά μέσο όρο 10%. Άρα σε ένα θεμελιώδες επίπεδο αναρωτιόμαστε, διαρωτόμαστε, θέλουμε να διευρύνουμε για άλλε δαπάνε έτσι υπέρ του αυστηρού όρου που ισχύουν για τι κρατικέ ενισχύσει, γιατί σε τελική ανάλυση πρέπει να προσέξουμε οι διατάξει να μην είναι πάρα πολύ περιοριστικέ. Πραγματικά για όλο το asset χρειαζόμαστε ένα κανονισμό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει παρέμβαση στα πλαίσια του asset ακόμα και αν, υπάρχει, αν δεν υπάρχουν απειλέ για την έννοια αγορά. Είναι ένα Πολύ θεμελιώδη σημείο αυτό, αλλά και σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο να το κοιτάξουμε αυτό δεδομένη και τη διάταξη ε, τη συνθήκη. Αν δεν υπάρξει πλήρη εναρμόνιση, το οποίο είναι απευκταίο, θα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε. Τρίτο ζήτημα, λοιπόν, πώ μπορούμε να εναρμονιστούμε με κοινού όρου, με συγκρίσιμα κριτήρια σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα. Στο σημείο λοιπόν αυτό Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πολύ πρόοδος ε, τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά για την απλοποίηση, για παράδειγμα, η εναλλακτική απλοποιημένου κόστους. Ίσως μπορούμε να εξηγήσουμε περισσότερο τα στοιχεία αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελούν μεγάλη απλοποίηση, μεγάλη βελτίωση. Να πω και το εξή. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις περιορισμένες όπου εξακολουθεί να υπάρχει κοινοποίηση. Δεν έχω τα επακριβή στατιστικά στοιχεία, αλλά θα μου έκανε έκπληξη αν είναι πάνω από 5 έως 10 κοινοποιήσει στη Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού ε, για τις δαπάνες ΕΣΥΦ ε, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά μέλος μπορεί να υπάρχει ένα περιστατικό κοινοποίησης ε, τα πέντε χρόνια, για παράδειγμα. Υπάρχει μια ανησυχία από πλευρά ε, τη πλευρά του ανταγωνισμού. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αναβάθμιση βιομηχανικού εξοπλισμού προκειμένου να τηρούνται τα κοινωτικά πρότυπα. Κάτι το οποίο επιτρέπεται από τα διευθυντικά ταμεία. Αλλά συνήθω δεν επιτρέψουν, δεν επιτρέπουμε στην κατοικία ενίσχυση να αναφερθεί σε τέτοια υποχρεωτικά πρότυπα για τον απλό λόγο ότι όλε οι εταιρείε ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινωτική αγορά θα πρέπει να πληρούν τους όρους αυτούς. Αν υπάρχει λοιπόν επιδότηση σε, κάποιους, ε, σε κάποιες εταιρείε, υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό καταδεικνύει ότι οι λίγες περιπτώσεις τις οποίες έχουμε μπορεί να μας πάρουν λίγο παραπάνω, γιατί αποτελούν προβλήματα ουσίας, ε, παρομοίως, κοινοποιήσεις για αμ, αυτοκινητοδρόμους που έχουν γίνει με εκχώρηση. Επί της αρχής δεν υπάρχει υποχρέωση κινητοποίηση γιατί δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση. Αν υπάρχει όμως εκχώρηση που είναι πιο παλιά και είναι λίγες εταιρείε εκχώρηση που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, είναι λίγοι όμιλοι και υπάρχει δυνατότητα μεγάλης υπέραποζημίωση όταν έχει γίνει άμα Μιλάμε όχι για 10 εκατομμύρια, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ασφαλώς και θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για την, τον ανταγωνισμό. Επίσης ε, και για τις κρατικές, ε, τα, κρατικά, τα, τα εθνικά δημοσιονομικά, αν υπάρχει υπερβολική αποζημίωση τέτοιων φορέων και οι ανταγωνιστέ ε, παρακολουθούν στενά τα ζητήματα αυτά. Αν δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι ανταγωνιστέ του ε, λαμβάνουν ε, κρατική ενέσχυση, προφανώ θα μα ζητήσουν να τα ερευνήσουμε αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν σε κάποιε περιπτώσει αυτά τα πράγματα παίρνουν πιο πολύ χρόνο για σωστού λόγου. Κάθε κράτο μέλο, ωστόσο, έχει ένα κέντρο των αρχών κρατικού, κρατικών ενισχύσεων. Ένα κέντρο συντονισμού που έχει και προνομιακές επαφές με, τις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγάλο ποσοστό γνώσης. Κάποια λοιπόν από τα θέματα τα οποία επισημάνθηκαν θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε σε πρώτη φάση. Για παράδειγμα, ο περιορισμός των τοπικών επενδύσεων, τα κέντρα επενδύσεων, η διάκριση δημοσίων ε, κοινών ε, εξόδων. Αλλά σήμερα θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους που μας παρουσίασαν λεπτομερέστατα και τους ευχαριστώ την κατάσταση στις χώρες της και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι από την άλλη Γενική Διεύθυνση ότι έτσι μπορούμε να εξετάσουμε πιο επισταμένους τα θέματα που μας παρουσιάσατε. Δεν θέλω να σας δώσω την εντύπωση σε καμία περίπτωση ότι είμαστε σε αμυντική θέση. Θέλουμε να σας ακούσουμε, θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι θέματα υπάρχουν και το τουλαχθέντος θα ήθελα να κάνω και κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τη φύση των δύο αυτών πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θα είστε σύντομος. Just to, flag as Να επισημάνω, όπως έχει ήδη γίνει, ότι εργαζόμαστε για την αύξηση του απλοποιημένου κόστους, γιατί εδώ έχουν ε, γίνει προτάσεις ε, βασικών πράξεων στα τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Και ο άλλος τομέας ε, όπου πραγματικά συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας είναι η εναρμόνιση του κόστους για τους ελέγχους και για την αξιολόγηση. Και πάλι λοιπόν θα χρειαστούμε αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει και ε, επαναχρησιμοποιούνται εφόσον είναι διαθέσιμες. Αυτό σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή στο νέο βασικό κανονισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόκληση, πρόσκληση. Ε, είμαι βεβαίως ότι θα αξιοποιήσετε την πρόσκληση αυτή και τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγητρία. Ναι, ναι. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Μπορεί να φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική τοποθέτηση μεταξύ των δύο θέσεων. Νομίζω ότι μπορούμε και με τις εκθέσεις και ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και με του συναδέλφους από την ΓΑΜΑΛΤΑ Ρέγκιο που εμείς εργαζόμαστε και από την Επιτροπή Μεταφορών εμείς έχουμε συνεργασία. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τι θέσεις αυτές. Είμαστε σε συνεχή διάλογο με την Κομισιόν, με τη ΓΑΜΑ Ανταγωνισμού, με τη ΓΑΜΑ Δέλτα για να βελτιώσουμε ακριβώ την κατάσταση, να μην υπάρχει αυτή η διπλή χρήση κτλ και η επικάλυψη. και να αξιοποιηθεί καλύτερα ο και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ξέρουμε ότι είναι πιο πολύ τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει και σωστός έλεγχος. Αλλά οι χώρες που, και οι αρχές που διαχειρίζεστε τις ενισχύσεις και έχετε σε επαφή με τους δικαιούχους, είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μιλήσατε για την αντίληψη που υπάρχει για το πόσο μπορεί να δοθεί προστιθέμενη, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά και τις πολιτικές εξαίρεσεις και τα λοιπά, κρατικές ενισχύσεις, ώστε να υπάρχει μια θετική αντίληψη επικοδομητική και από τις Ευρωπαϊκές Πόλεις και από τις εθνικές διοικήσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ. Κάθε φορά που προσπαθούμε να βελτιώσουμε ή να πλουστεύσουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό ή κάθε φορά που προσπαθούμε στους προσεχείς προϋπολογισμούς ε, ή στην απαλλαγή να εντάξουμε κάποιες συστάσεις και υποδείξεις ε, που ακριβώς στόχο έχουν την απλούστευση. Γιατί ανησυχούμε με το ότι αυξάνεται η εντύπωση ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι τόσο πια πολύπλοκος ε, ιδίως ό,τι αφορά δυνατότητε παροχή παροχής βοήθειας, είναι τόσο δύσκολο να γίνουν κατανοητοί κανόνες, ώστε να ζητούνται άλλες αναλλακτικέ τελικά. Και η έλλειψη πραγματικότητα μας ανισχύει και εμάς. Όσα είπατε λοιπόν θα τα μεταφέρουμε στους εκπροσώπους της Κομισιόν, που είναι και αυτοί οι οποίοι παρουσίασαν μια δεσμέτρων που θα μελετήσουμε ενδελεχώς για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις για τα θέματα που θέσετε επιτάπητος. Υπάρχουν διαφορετικοί σκοποί και στόχοι τόποι Κομισιόν, άρα θα είναι δύσκολο ίσως να συμφιλειωθούν ε, πάντοτε αυτοί οι διαφορετικοί στόχοι. Το θέμα είναι να βρούμε τον κατάλληλο ορισμό, ίσως ένα διαφορετικό ορισμό, που να μην ε, δημιουργεί και αντιφάσεις όμως. Νομίζω λίγο πολύ αυτό είναι το μήνυμα που μας ε, δώσατε και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσπάθεια που κάνετε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ε, και το διάλογο μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να δισκεδάσουμε τις ανησυχίες σας εν τέλει. Ευχαριστώ. Um, uh, σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να πω κάτι. πιο παρατηρητικοί θα δουν ότι θα έχουν παρατηρήσει ότι δεν είμαι η κυρία Γκρέσλε. Ε, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, αλλά και εγώ δυστυχώς ε, πρέπει να πάω σε μια άλλη επιτροπή ε, που πρέπει να είμαι εκεί στις 5. Θα δώσω λοιπόν την προεδρία στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα είστε εισηγήτρια και πρόεδρος ταυτόχρονα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Ευχαριστώ. Derek. Ε, Ωραία, λοιπόν, τότε θα περάσουμε. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν το λόγο, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που έχει να κάνει με το πώς θα ενημερώσουμε και θα βελτιώσουμε την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Με το, τον κύριο Μπροκόπ από το ενεκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτήν την ακρόαση και δεύτερον θα ήθελα να πω ότι ε, θέλουμε να δούμε αν είναι συγκρίσιμα αυτά τα ε, συζητήματα. Έχουμε την ειδική έκθεση του 16. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να ε, υπάρξει ενημέρωση και να υπάρξει η ε, ευθυγράμμιση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Τα στοιχεία που έχουμε είναι από το 2016 και από το 2017. Στην δική μας έκθεση εξετάσαμε τα σφάλματα που σχετίζονταν με το οικονομικό έτος 2014. Βρήκαμε 15 περιπτώσεις ε, 13,5 του ετησίου ε, σφάλματος. Ε, μεγάλο τμήμα δε ε, σχετιζόταν με το, τα διευθυντικά ταμεία και την, το ΣΕΦ, δηλαδή το Ταμείο Συνοχής. συχνά αυτά ε, εμπίπτουν στον κανόνα ντεμίνιμις και άρα δεν είναι εύκολο να υπάρξουν εκεί λάθη. Έχουμε ταξινομήσει τα σφάλματα σε τέσσερις κατηγορίες. Αυτά που είναι τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά όπου έχουμε ε, οικονομικό αντίκτυπο και έχουμε πέντε ε, σφάλματα όσον αφορά ε, την ε, κατηγορία αυτή των ε, σφαλμάτων. Επίσης εξετάσαμε τα θέματα μη συμμόρφωσης και αναλύσαμε αυτά που βρέθηκαν. Προσπαθούσαμε να δούμε τι έκανε η Κομισιόν ή τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ανέβρεση αυτών των σφαλμάτων. Η DG Regio και η EMCO βρήκαν σφάλματα και, και εντόπισαν διάφορα προβληματικά προγράμματα ενισχύσεων. Είδαμε πως η Κομισιόν είχε καταγράψει τα σφάλματα στα συστήματά της, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει συνολική ανάλυση για να δει κατά πόσο ε, επαναλήφθηκαν ή όχι αυτά τα σφάλματα. Σε σχέση με τα σφάλματα είδαμε ότι η DG Regio επέβαλε οικονομικές διορθώσεις, αλλά ότι δεν έγιναν σημαντικές ανακτήσεις από την DG Comp. Επίσης διαπιστώσαμε για τους εξάντε όρους για την περίοδο 2014 πως ήταν θετική αλλά ότι ορισμένα κράτη-μέλη στην, ε, κατά τον έλεγχο φάνηκε να έχουν προβλήματα που δεν συνέπεπταν με την εκτίμηση. Ένα σημαντικό θέμα είναι, όπως ανέφεραν και κάποιοι άλλοι ομιλητές, ήταν τα στοιχεία του GBED, όπου έχουμε ε, μία εκτίμηση για το σφάλμα, ε, το οποίο θα δείτε στην διαφάνεια τα μέτρα που καλύπτονται από το Deeper το 2014 όπως είπε και ο κύριος Κόπμαν, είδαμε ότι έχουμε φτάσει σε κάλυψη 90% και με τις δαπάνες φτάσαμε στα 2 τρίτα που καλύπτονται και πάλι εκεί ε, φτάνουμε στο 74%. Σημαντικές αλλαγές ήταν η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, αλλά υπήρχε και αλλαγή στην εφαρμογή του αρχικού κινήτρου. Αυτό θα δείτε ότι είναι σημαντικό και σε σχέση με την ε, ανέβρεση ζητημάτων μη συμμόρφωσης. Για τα έτη 2010 μέχρι 2014 έχουμε βγάλει τα πορίσματά μας από τις αιτήσει εκθέσεις του 2015 και του 2016 και έχουμε τα εξή να πούμε. Είδαμε ότι ξεκολουθούσε να υπάρχει κάποια μη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, αλλά φαίνεται να έχουμε λιγότερα σφάλματα με οικονομικό αντίκτυπο. έχουμε και την αναδρομική εφαρμογή του κανονισμού σε συγκεκριμένα πορίσματα. Για το 2015 βρήκαμε 7 περιπτώσεις και στο 2016 11 υποθέσεις, αλλά χωρίς φάλματα με, οικονομική, ε, με οικονομικό αντίκτυπο. Στην ειδική έκθεση Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και κάποιες καλές πρακτικές. Ο, μία σχετίζεται με τη γενική διαδικασία που ασχολείται με όλα τα ε, project. Πρόκειται για κρατική, ε, κρατικό έλεγχο όλων των νομοθετικών προτάσεων που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη φάση. Μια άλλη καλή πρακτική που τονίσαμε ήταν από την Πορτογαλία που ήταν πιο εστιασμένη ε, σε σχέση με τα, τα ανώτατα όρια de όπου υπήρχε ένας κεντρικός κατάλογος για τα de Είδαμε από τις κρατικές ε, ε, αρχές ελέγχου πως βλέπουν το θέμα αυτό είναι αρκετά δύσκολο, περίπλοκο μάλλον, ή πολύ περίπλοκο και γι' αυτό είπαν ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένας οδηγός, ε, πρακτικές, ε, ε, πρακτικά παραδείγματα. Έχει υπάρξει επίσης ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο έχει φτιάξει DG Radio με την DG Coma. Αυτό από ό,τι ακούσαμε από τους συναδέλφους της Επιτροπής έχει ενημερωθεί αρκετές φορές. Το τελευταίο καλύπτει την περίοδο 2018 μέχρι 2020 ε, και για να ενισχυθεί η εφαρμογή, το συστήναμε και στην έκθεσή μας, η Κομισιόν θα πρέπει να καταγράφει τις παρατεπίες που διαπιστώνει και να μπορέσει έτσι να κάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση και σε σχέση με το, τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει πως η έλεγχοι των αρχών είναι σωστή, δίνουν επιπλέον κατευθύνες γραμμές και ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να ορίζουν ένα συγκεκριμένο κατάλογο όσον αφορά τις δεμήνυμες ενισχύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόκοπ. Μας κάνατε κάποιες πενθυμίσεις και σας ευχαριστώ όπως και για την προσπάθεια να μας θυμίσετε τι έχει κάνει ήδη το ελεγκτικό συνέδριο. Και ξέρουμε και ότι η Κομισιόν έχει καταθέσει νέες προτάσεις ε, που ελπίζουμε πως πηγαίνουν στην διακατεύθυνση. Ο κύριος Λόι Βάγνερ τώρα. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να μας πει τις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ορίστε. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Κύριε Φερνάντες, είχε ζητήσει το λόγο. Ναι. Για την παρουσίαση του Ανθρωπικού Συνεδρίου είχα κάποια παρατήρηση. Οι συστάσεις προς τη ΔΕΛΤΑ ΡΕΓΚΙΟ έχουν εφαρμοστεί. Η πρώτη σύσταση με το σχέδιο δράσης ε, για καθεύτηρες γραμμές και εκπαίδευση στα κρατημέλη. Σε ό,τι αφορά το Μητρό Παρατυπιών, καταγράφουμε τα πορίσματά μας ε, και από φέτος προσθέτουμε στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την τυπολογία των ασφαλμάτων που εντόπισαν ελεκτικές αρχές και τρίτον δίνουμε καθοδήγηση στις ελεκτικές αρχές. Το είπα και στην παρουσίασή μου. Γιατί τους μεταφέρουμε το checklist και τους ζητούμε να χρησιμοποιούν όλοι οι ελεκτέ από όλες τις χώρες το ίδιο checklist. Σας ευχαριστούμε. Ναι, ήμουν βεβαίω ότι είχε υπάρξει ήδη βελτίωση. Γιατί πέρασε και κάποιο καιρό από τότε που δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο πριν δώσω στον επόμενο μιλητή. Τον τελευταίο για σήμερα, τον κύριο Λόικ Βάγκνερ, όπω είπα, από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Να μα πει λοιπόν ποιε είναι οι διαδικασίε. σε ό,τι αφορά το δικαστήριο. Πού είστε κύριε Βάγνερ? Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγήτρια, εξωτικού βουλευτέ. Θέλω να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ακρόαση με θέμα κρατικέ ενισχύσει και χρηματοδότηση ένωση, αν είναι συμβατά αυτά τα δύο μεταξύ του. Σημαντικέ επιτυχίε οικονομικέ, χρηματοπιστωτικέ, πολιτικέ, νομικέ. σε ό,τι αφορά τον ε, δικαστικό και νομικό έλεγχο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές δικαστικές ε, διαμάχες από το 2010. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα μπορούμε να δούμε τι γίνεται από τις κρατικές ενισχύσεις. Για την περίοδο 54 έως 2009 ήταν λιγότερες υποθέσεις από ό,τι για αυτή την περίοδο από το 2010 και μετά. ποια είναι τα θέματα και υποθέσεις. Δεν έχουμε μονοκρατικές ενισχύσεις, αλλά και διαθωτικά ταμεία και βλέπουμε το αποτέλεσμα που είναι πολύ σημαντικό. Μειώνονται οι υποθέσεις. Υπάρχουν και κάποιες προσφυγές ε, ακύρωσης που δεν κρίθηκαν παραδεκτές. Βγάζουμε λοιπόν τις μη παραδεκτές υποθέσεις, άρα μειώνεται ακόμη περισσότερο. Μένουν τρεις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με κρατικέ ενισχύσεις ε, και πολιτική, οικονομική κοινωνική εδαφική συνοχή. Το δικαστήριο σπάνια εκλήθη να συζητήσει για το πώς σχετίζονται οι κρατικές ενισχύσεις με τα διαρθρωτικά ταμεία. Μόνο εάν μας προσκαλέσουν οι διάδικοι μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Και το είπαμε και σε μια απόφαση στη... κατά τον κόντρα η Dynamics. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε όλοι τραπετίτα. Εγώ θα εστιάσω στον δικαστικό έλεγχο. Στην έννοια κρατικών πόρων με βάση το άθρο 107 για τη διάρθρωση της κοινωνικής πολιτικής και των κρατικών ενισχύσεων και τις κρατικές ενισχύσεις και την οικονομική, πολιτική, και κοινωνική συνοχή. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, το νομικό και την, ε, το πεδίο εφαρμογή του. Θέλουμε να υπάρχει ε, ένας, ε, μια ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν, κατά περίπτωση, ασκούμε ή περιορισμένο ή πλήρη έλεγχο για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν σήμερα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ε, από ε, την ουσία θα είμαι πολύ σχηματικός λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ε, σε ό,τι αφορά αν χαρακτηρίζεται κρατική ενίσχυση ανάμεσα του άρθρου 107, θεωρούμε ότι υπάρχει έλεγχος και πρέπει να είναι αυτός πλήρης που θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα ή μη συμβατότητα ενός μέτρου ενίσχυσης, πάντα θεωρούσαμε από το 80 ήδη ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι τέτοιο. 27 Φεβρουαρίου του 2014 στην υπόθεση Ακανφόρα το δικαστήριο λέει ότι δεν είναι ψηλωσίας αρμόδιο για να αποφασίσει ένα προδικαστικό ερώτημα για την ε, συμβατότητα τη κρατική βοήθειας. Εφαρμογή παρεκκλήσεων από το άρθρο 107 παράγραφος 3. Μιλάω για τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ένωση. Με βάση σταθερή νομολογία έχει η Κομισιόν ε, τη δυνατότητα τη διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. στο πλαίσιο πολιτικών όπως η πολιτική συνοχή, πάντα κατασταθερή πάγια ομολογία. Στην υπόθεση Πολωνία κατά Κομισιόν, ο έλεγχος του δικαστήριου είναι περιορισμένος, γιατί δεν είναι δική μας αρμοδιότητα το θέμα άρθρο 107 Συνδίκη για τη λειτουργία της Ένωσης και η απέτηση κραστικού πόρου. Χεσόχ Ντετά. 9 Ιουνίου του 82 ε, για το Βόλιο Κρέας. Είχαμε προδικαστικό ερώτημα για τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν ε, την δασμολογική ποσόστοση για το βόλιο κρέας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε αυτή την υπόθεση κρίναμε ότι τα μέτρα περιορίζονται στην κατανομή της ε, ε, ποσόστοσης δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Το χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα δεν δίνεται μέσω κρατικού πόρου, αλλά κοινοτικού πόρου. Alors, par la Σλόμα Νεπτούν, 93, νομολογία του δικαστηρίου. Και εκεί ξεκάθαρα λέμε ότι υπάρχει μια διάκριση στις συνθήκες. Ενίσχυση που δίνεται μέσω κρατικών πόρων ή ενίσχυση από κράτη-μέλη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις που δίνονται από το κράτος ή από οργανισμούς που έχουν οριστεί ή σχεδιαστεί από το κράτος. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Πρόσφατα, 9 Νοεμβρίου 17, απόφαση Κομισιόν έναντι TV2 Δανία. Θυμίζουμε ότι περιλαμβάνεται σε τίσχες, στις κρατικές ενισχύσεις και αυτές που δίνονται από ενδιάμεσους. Κρατική πόρη είναι όλα τα πόσα, τα οποία είναι υπό δημόσιο έλεγχο και άρα στη διάρκεια των εθνικών αρχών, ακόμη και αν δεν είναι μονίμως στα δημόσια ταμεία αυτά τα κονδύλια. Ακυρώνει έτσι απόφαση του δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είχε ερμηνεύσει περιοριστικά τον όρο κρατική πόρη. Ressources d'État. Ξεκαθαρίσαμε και το θέμα των κρατικών πόρων. Τώρα, τα διευθυντικά ταμεία πολλές φορές έχουν και ένα άλλο, μια άλλη πτυχή, το γεωργικό ταμείο, ΦΕΝΤΕΡ και ΦΕΟΓΑ. Άρα θα αναφερθώ τώρα στις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Άρθρο 42 της Συνθήκης Εκλήτησης λέει ότι οι διατάξει του κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και διάθεση στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων στο μέτρο που ορίζεται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Ποιε είναι οι επιπτώσει αυτών των διατάξεων σε ό,τι αφορά των αρχιτεκτονικών ενισχύσεων. Έχουμε μια απόφαση τη Δευτέρα Δεκεμβρίου του 10. Βολάνε το Μάλτ κατά τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ένα παράδειγμα. Έχουμε απόφαση της Κομισιόν ως βάση. Για μια στοπία. Υποτίθεται ότι έπρεπε να υπήρχαν ε, κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες, ε, οι οποίες περιλαμβάνοντας κατευθύνσεις γραμμές για την κοινωνική πολιτική. Το δικαστήριο δηλώνει ότι περτερεί η κοινή γεωργική πολιτική στους στόχους ε, της πολιτικής ανταγωνισμού. Ε, πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής. Έπρεπε η Κομισιόν να λάβει υπόψη τον έλεγχο της παραγωγής. Όπως προέβλεπαν τότε διατάξεις, φεογκά, ταμείο προσανατολισμού στόχο αύξηση παραγωγής ε, προϊόντων που δεν έχουν ε, εύκολη πρόσβαση στις αγορές. Αλλά δεν ήταν συμβατή κατά το δικαστήριο αυτή η κρατική ενίσχυση που αύξησε την παραγωγή του προϊόντος, αυτό που δεν θα μπορούσε όμως να διατεθεί ε, στην αγορά και να ωφελήσει και την περιοχή. Και έρχομαι τώρα σε κάποιες άλλες υποθέσει του δικαστηρίου για κρατικές ενισχύσει και την πολιτική κοινωνική οικονομική συνοχή. Σας έλεγα ότι έχουμε τρει τέτοιε υποθέσει ουσιαστικά επί τη ουσίας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη αφορά πολιτική συνοχή και δικαίωμα κρατικών ενισχύσεων. Οι άλλε δύο πιο τεχνικέ. Θα προσπαθήσω να τι απλουστεύσω στο μέτρο του δυνατού εφόσον βασίζονται σε προηγούμενες διατάξεις από το 99. Σε απόφαση 8 Νοεμβρίου 2008, Χοτέλ Σιπριάνη και άλλοι κατά της Κομισιόν, το δικαστήριο εκτιμά ότι σωστά η Κομισιόν θεωρεί του πολιτική ανταγωνισμού και συνοχή κοινωνική οικονομική κτλ. Είναι δύο διαφορετικέ, αυτόνομε πολιτικέ. Τα διαφορετικά ταμεία λοιπόν είναι το βασικό μέσο της πολιτικής Συνοχή και η εξαίρεση του 107 για τις περιφερειακές ενισχύσεις εμπίπτει στην πολιτική ανταγωνισμού. Και ουσιαστικά απλά αποφεύγει τις τρευλώσει. Σε αυτή την υπόφαση λοιπόν λέει το δικαστήριο ότι είναι συμπληρωματικέ ό,τι αφορά περιφερειακέ περιφερειακές ενισχύσεις δύο αλλά δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ των στόχων των δύο πολιτικών. Δηλαδή, οι στόχοι οικονομική ε, πολιτική συνοχή δεν είναι κάτι που υπερτερεί των στόχων τη πολιτική ανταγωνισμού, ούτε και το αντίθετο. Η Κομισιόν λοιπόν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζει πιο ευέλικτα ε, τις αρχές ανταγωνισμού για προς όφελος των στόχων της πολιτικής συνοχής. Και ήδη τότε είχαμε πει ότι οι καθεντρίες γραμμές του 98 περίχαν ειδικέ διατάξεις υπέρ της ε, μεγαλύτερης συνεκτικότητας των κανόνων και βέβαια όριζαν συγκεκριμένου κανόνες για τον ανταγωνισμό. 9 Ιουνίου του 2011 έχουμε μια απόφαση του δικαστήριου. Κομιτά το Βενέτσια, Βόλε, Βίβερε κλπ. κατά της Κομισιόν. Δεν εξεφράστη το δικαστήριο προς το παρόν. Μια άλλη υπόθεση τώρα. Celle du 24 novembre 2005, Italie contre Commission. 24 Νοεμβρίου του 2005, Ιταλία κατά Κομισιόν. Α, με συγχωρείτε, λάθος. Δεν είναι το πρωτοβάθμιο, αλλά το δικαστήριο το ευρωπαϊκό που την έχει βγάλει αυτή την απόφαση. Εδώ είχαμε κάποια προβλήματα επιλεξιμότητας κάποιων προκαταβολών που είχαν δοθεί σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσει. Ότι δηλαδή δεν είχαν κατατεθεί παραστατικά ή τέλο πάντων άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω δαπάνε ε, είχαν χρηματοδοτήσει στόχου που καλύπτονται από τα διορθωτικά ταμεία. Δημοκρατία θεωρούσε ότι καμία διάταξη, ούτε ο Γενικός Κανονισμός, ε, ούτε ούτε οι εφαρμοστικές διατάξεις επέτρεπαν να θεωρηθεί ότι θα έπρεπε να επαληθευτεί η δραστηριότητα των δικαιούχων, των τελικών δικαιούχων όπως λέγονται. Απερίφθη από το, το Δικαστήριο αυτή η υπόθεση, αυτή η αίτηση ακύρωσης. Ένας από τους στόχους, λέγεται από το δικαστήριο, είναι να υπάρχουν εγγυήσεις χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι δαπάνες. Βέβαια, η απόφαση τα λέει πολύ πιο λεπτομεριακά. Επί της ουσίας όμως θεωρεί το δικαστήριο ότι μπορεί να απαιτεί τα παραστατικά αυτά η Κομισιόν τελικά και για τις ενδιάμεσες πληρωμές και για την εξώσφυλση του υπολείπου. Αυτά πάντα για τον προηγούμενο κανονισμό. Μάλλον ξεπέρασα το χρόνο μου, οπότε να μην μιλήσω για τις 12 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση Ιταλία κατά την Κομισιό ΤΙΦ 308 κάθετος 05. Λίγο πολύ περί της ίδιας υπόθεσης πρόκειται. Απλά εκεί τροποποιείται η διάταξη Εκεί το θέμα ήταν ε, κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Παραβίαση αρχή ίση μεταχείρισης, είπε η Ιταλία, δεν συμφώνησε το δικαστήριο. Με βάση τα επιχειρήματα της Κομισιόν και την ανάλυση ε, αυτή ε, πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, άρα διαφορετική και μεταχείριση, λέει το δικαστήριο. Στην περίπτωση επιχειρηματικού κινδύνου είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος. Μια πρόσφατη υπόθεση. Υπόφαση Μην ανησυχείτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα περιοριστώ σε αυτά που μας ενδιαφέρουν μόνο. Να σας πω ποια ήταν τα πραγματικά περιστατικά. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, το ξέρουμε. Γιατί συνδέεται με τη σημερινή θεματολογία. Όμως, από νομικής πλευράς, το θέμα ήταν αποκλειστικά ο γενικός κανονισμός εξαίρεσης ανακατηγορία το 2008 και δεν, λαμβάνει, ε, δεν αποφασίζει επί άλλων θεμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας τα είπατε πολύ νομικά τα πράγματα. Ε, ίσως ένα κομμάτι να το καταλάβαμε ενδεχομένω. Θα ήθελε κάποιο το λόγο, από την Κομισιόν ίσως, ή κάποιος άλλος, για να απαντήσει Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος. Και δεν υπάρχουν και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και θα τα μελετήσουμε ενδελεχέστατα. Όσα μας είπατε και τις παρουσιάσεις της άλλες θα τις μελετήσουμε. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, θέλουμε να προετοιμαστούμε, ώστε το δυνατόν καλύτερα. Γιατί έπεται συζήτηση σε σχέση, σε σχέση λέω, με το νέο προπολογισμό για μετά το 20. Ακούσαμε την άποψη των πόλων, των, περιοχών, μάλλον των περιφερειών, των κρατών, των δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, άμεσες ενισχύσεις και τη ρύθμιση σχετικά, πώς την κρίνουν γενικώ. Στόχος είναι να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο για όλους τους κοινωνικονομικούς ε, φορείς που εργάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν και ο στόχος ακρόασή μας, να καταλάβουμε τι γίνεται. να ακούσουμε όλες τις πτυχές, να δούμε τι βελτιώσεις έχουν γίνει, να θέσουμε τις ερωτήσεις μας, να ακούσουμε τι λένε οι διοικήσεις και τι λένε οι δικαιούχοι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν ακόμη και πρέπει να τεθούν για να βρεθούν λύσεις. Και τέλος, βεβαίως, έχουμε τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου που εντοπίζουν ε, πώς να το πω, ε, κάποιες ανησυχίες, ε, κάποια σφάλματα για συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται ε, της ιεράρχησης, τη συμπληρωματικότητας που μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει σε ό,τι αφορά τις μορφές ενίσχυσης και τις διάφορες πολιτικές δίκαιου ανταγωνισμού. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ορισμένα μείζωνα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε για να ε, καταλήξουμε σε έναν δίκαιο και επαρκή ε, για να καλύψει τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό προπολογισμό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλες αυτές τις πληροφορίες και θα είμαστε σε επαφή μαζί σας, σίγουρα με την Κομισιόν. Θα εμβαθύνουμε και σε κάποια ερωτήματα, σε κάποια στοιχεία που πρέπει να μελετήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα. Είναι διαφορετικέ οι δύο πολιτικέ, τέλο πάντων έχουν διαφορετικού στόχου. Αλήθεια είναι αυτό, όμω ο τελικό στόχο, ο απότατο στόχο, ποιο είναι. Οι οικονομικέ και κοινωνικέ πολιτικέ της Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό τον προπολογισμό να προσφέρουν τα, δυνατό, τα μεγάλα δυνατά ωφέλη. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Τα σημειώσαμε όλα. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά είχαμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε ορισμένα ζητήματα και ελπίζω και στο μέλλον να μπορούμε να διατυπώσουμε τα σωστά ερωτήματα σε όλου ε, του εμπλεκόμενου φορεί για τον νέο προπολογισμό και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε και την εφαρμογή του και τον έλεγχο. Αυτή είναι η στόχη τη δική μα επιτροπή, όπω γνωρίζετε πολύ καλά. Σα ευχαριστώ. Και θα περάσω στο επόμενο σημείο τη μερική διάταξη. Sí. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, που είναι η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου 14-2018 και που επίσης περιλαμβανόταν στην απαλλαγή για το 2017 και αφορά τα κέντρα αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά όπου το ελεκτικό συνέδριο μας λέει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος. Η κυρία Γιάκομψένα, το ελεκτικό συνέδριο, θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για την χημικά, την πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστεία, για χημικά και βιολογικά και ραδιολογικά. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν αποτελεί ένα βασικό πρόγραμμα για την ελαχιστοποίηση τέτοιων απειλών και κινδύνων από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι κίνδυνοι λοιπόν ε, αποτελούν σημαντική απειλή για την υγεία, για το περιβάλλον και για την οικονομία. από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ε, διαχειριζόμαστε την ε, πρωτοβουλία αυτή για 139 ε, εκατομμύρια ευρώ και για την περίοδο 2014-2020 130 εκατομμύρια ευρώ. Και σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την ικανότητα των υπεύθυνων αρχών για την αντιμετώπιση των απειλών ΣΥΠΙΑ και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ε, αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών αρχών. Ο Στόχο ε, του ελέγχου μα λοιπόν ήταν διτός. Καταρχάς να παρακολουθήσουμε και να καταμετρήσουμε τι ε, δράσει τη ΙΕΕΣ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνουμε να δούμε κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί οι συστάσεις του 2014 της προηγούμενης έκθεσης σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία αυτή και κατά δεύτερον να αξιολογηθεί κατά πόσο η πρωτοβουλία έχει συμβάλει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση και μείωση των χημικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρακολουθήσαμε και εξετάσαμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν εφαρμόσει μια σωστή στρατηγική για την διαχείριση κινδύνων, κατά πόσο η πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί επαρκώς και ικανοποιητικώς στις χώρες εταίρους και κατά πόσον η σωστή παρακολουθήση και τα συστήματα αξιολόγησης έχουν συσταθεί για την αξιολόγηση και παρακολούθηση και υποβολή αναφορών των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας. Το συμπέρασμα στην έκθεσή μας είναι ότι η πρωτοβουλία όντως έχει ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους CPI, αλλά παραμένουν πολύ κίνδυνοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Δράσης έχουν εφαρμόσει τρία Τρεις από τις έξι συστάσεις που περιλαμβάνονται και στην προηγούμενη δική μας έκθεση και εφαρμόζονται μερικώ σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η σύσταση για την επικέντρωση της Ευρωπαϊκής ε, χρηματοδότηση στους πιο απαραίτητους τομείς ε, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και πιστεύουμε ότι η σωστή και κατάλληλη προσέγγιση για τη χρήση κινδύνων δεν έχει αναπτυχθεί στο έπακρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στις χώρες εταίρους ε, εργαλεία μια μεθοδολογία προκειμένου να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους CPI. Ωστόσο, η καθοδήγηση για το πώς θα εντοπίζεται ο κίνδυνος και πώς θα ιεραρχείται ο κίνδυνος θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνεται να απαντήσει αρκετά εγκαίρως στα αιτήματα ρογής από τις χώρες εταιρού, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη συνεργασία και τις εθνικές ομάδες CPI που έχουν οριστεί στην πλειονότητα των κρατών αυτών τα έργα θεωρούμε ότι έχουν πετύχει τα πιο πολλά αποτελέσματά τους και οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, συμμετέχουν στην ανάπτυξη δυναμικού. Ωστόσο, η περιφερειακή συνεργασία ακόμα ύστερη. Έχει βελτιωθεί μεν η συμμετοχή της ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι επαρκώς ενεργή και δραστήρια για να προωθήσει την όλη πρωτοβουλία και την ε, διάδραση μεταξύ των Γενικών Διευθυνσέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κοινότητα των δωρετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί, αξιολογεί, αλλά δεν υπάρχει α, σωστός καθορισμός των ενδεικτών των προτεραιοτήτων και αυτό καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση του αντικτύπου τι συστήνουμε λοιπόν, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την πρωτοβουλία αυτή, συστήνουμε η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ιεραρχήσουν σωστά τι δραστηριότητε βάση ε, αξιολόγηση συστημικού κινδύνου, να ενισχύσουν ε, την περιφερειακή διάσταση της πρωτοβουλία, να ε, ενισχύσουν περαιτέρω τη αντιπροσωπεία και τη συμμετοχή τη αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοβουλία να εντοπίσουν σωστέ ε, πηγές χρηματοδότηση να τονίσουν την ε, προβολή και την διαφάνεια των διαδικασιών αυτών σε ό,τι αφορά και την αξιολόγηση και τέλος ε, να επιτρέψουν εύκολη πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε που σχετίζονται με την πρωτοβουλία Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν αποδεκτεί και τι έξι αυτέ τι τάσει τη εκθέσει μα και θα ήθελα να του ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία του κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγή του ελέγχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κόμψεν. Εγώ εξ ονόματος τη ομάδα μου πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του κύριου Μπαλσίτη του εισηγητή. Και θα ήθελα να σας ε, διαβιβάσω την γνώμη του. Καταρχάς αναγνωρίζει πως ε, η έκθεση αυτή μας δίνει ένα γενικό ευρύ πανόραμα για τις δραστηριότητες αυτών των κέντρων. Συμφωνεί με τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και με τις συστάσεις του και θα ήθελε μόνο να προσθέσει δύο σχόλια. Καταρχάς, την ανάγκη για ενίσχυση της ε, περιφερειακής διάστασης της πρωτοβουλίας. Σύσταση παριθμών 2 και το γεγονός ότι η περιφερειακή συνεργασία έχει σημασία για να εντοπιστούν κοινοί στόχοι, αλλά και έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτής της πρωτοβουλίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μεγαλύτερης συνοχής και συνέπειας ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές ε, που εφαρμόζονται στις ε, χώρες εταίρους. Εδώ μιλάμε για κέντρα αριστείας και θα πρέπει αυτή η πολιτική να ενταχθεί στο ε, πρόγραμμα το πολιτικό για να μπορέσει να βελτιωθεί η συνέπεια και να ενισχυθεί η συνεργασία. Εγώ θα ήθελα όλος ιδιαίτερος να αναφερθώ στο γεγονός ότι η δικαιολόγηση, η εξήγηση που δίνει η Κομισιόν σε σχέση με τις ε, δυσκολίες μιας πιο περιφερειακής προσέγγισης ή σε σχέση με μια τοποθέτηση γενικότερη, εγώ κατανοώ από πλευρά της Κομισιόν ότι υπήρξε μια διεύρυνση και ότι κάθε φορά χρειαζόμαστε περισσότερο γιατί είναι απαραίτητο οι χώρες των διαφόρων περιφερειών να μπορέσουν να ε, υιοθετήσουν αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούν ε, επί των κινδύνων που είναι κάθε φορά μεγαλύτεροι σε σχέση με συγκεκριμένα πλαίσια περιφερειακά. Να αναγνωρίζω γιατί εγώ ασχολούμαι και με το Μαγκρέμπ πως είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε και τις σχέσεις ε, ανάμεσα στις διάφορες χώρες και την κατάστασή τους που πώς και κατά πόσο έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και τέλος αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, την κυρία Γιάκομψεν είναι αν εσείς προσέξατε αυτήν την ενημέρωση που υπάρχει από το προσωπικό που εργάστηκε σε αυτή την πρωτοβουλία φαίνεται να μειώθηκε κατά 50%. Μου φαίνεται τεράστιο. Μια τέτοια σπουδαία πρωτοβουλία να έχει περικοπεί τόσο δραστικά το προσωπικό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το λάβατε υπόψη. Όταν συντάσσετε τις συστάσεις σας, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε ε, για αυτό το έτος, το 2017, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις για το μέλλον θα πρέπει να λάβουν περισσότερη υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δουλέψει περισσότερο με αυτά τα κράτη. Σας ευχαριστώ. Sí, perdone, sí, ναι, συγγνώμη κύριε Γιάκοψεν. Ε, ε, αν δεν σας πειράζει να δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Έντι Μάγερ. Παρακαλώ. που είναι επικεφαλής της Ντέζε Ντεύκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πάντα ήταν καλή συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο. Ήταν πραγματικά χαρά μα που συνεργαστήκαμε μαζί του και μα βοήθησαν ιδιαίτερα. Γιατί φαντάζεστε ότι μια πρωτοβουλία τέτοιου επίπεδου που ξεκίνησε από το 0 του 2011 ήταν μια σαφή και μόνο ιδέα πλέον έχει πραγματοποιηθεί και έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία με 60 χώρες σε 8 περιοχές εταιρείε οι οποίε πρόσφατα προσχώρησαν Αφγανιστάν, Πακιστάν και που ασφαλώς βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση ω προς την ασφάλεια και αποδέχτηκαν να συζητήσουν θέματα ασφάλειας μαζί μας για όλη την περιοχή. Και μόνο γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι περήφανη που το πέτυχε αυτό. Σα ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι για τη βοήθειά σα. Ε, και ναι, για το τελευταίο σχόλιο σας. Ε. Και εμείς ε, έχουμε περικοπές προσωπικού όπως και άλλες ε, υπηρεσίες από την Επιτροπή. Και κυρίως αυτό έπληξε τους ε, συναδέλφους από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για διάφορες χώρες. Αυτό προφανώς έχει επιβραδύνει τις ικανότητές μας. Και θα πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε να βάζουμε κάποια τάξη στην όλη κατάσταση. Το κέντρο αριστεία είναι ένα πολύ περίπλοκο οικοδομήμα από την αρχή. Ήταν πολύ φιλόδοξο ο στόχος και κάλυψε καταρχάς φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, τρομοκρατικού τύπου ζητήματα και το CBRN εκρηκτικά, κυβερνοέγκλημα πλέον ως στόχο του κέντρου. Είναι πολύ ευρύ λοιπόν το πεδίο και αυτό αντικαταπτρίζει και αυτά που αντιμετωπίζουμε άλλωστε καθημερινά. Καθημερινά στον κόσμο σε ό,τι αφορά του κινδύνου δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια μικρή συζήτηση μεταξύ ημών και του ελεγκτικού συνεδρίου για το πώς θα χαρακτηριστούμε, πώς θα επιλέξουμε τον τύπο κινδύνου που εφαρμόζουμε. Καταρχάς, επαφείται στις χώρες εταίρους να αποφασίσουν ε, πού θέλουν να συνεργαστούν και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα από τα σημεία επιτυχίας ε, του κέντρου αριστείας. Δεν επιβάλλουμε τίποτα. τα κράτη το συζητούν σε επίπεδο επιτροπή, σε επίπεδο περιφερειακό και εθνικό για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Και φυσικά αυτό δεν συνάδει απόλυτα πάντα με τους ε, κίνδυνου και τι προτεραιότητες τη Ένωση. Και επιπροσθέτω, ο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άμεση γείτονες μας. Ε, Βόρειο Αφρική, Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική από την οποία κυρίως προέρχονται οι τρομοκρατικέ απειλές, αλλά έχουμε και άλλους κινδύνου του οποίους του ξεχνάμε κατά καιρού. Οι αγρότε μας μας τα υπενθυμίζουν σε ό,τι αφορά παράδειγμα την γρήπη των πτηνών από την ε, Ασία που έπλεξε σημαντικό τμήμα των πτηνών και προκάλεσε μεγάλες ζημίες στην οικονομία μας θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συνδεθούμε μόνο με τους ανθρώπους γιατί η οικονομία αντιμετωπίζει και άλλες επιθέσεις πολύ σημαντικές και αυτό ο ιστορικός πώς εξηγεί γιατί η Νοτιοανατολική Ασία είναι πιο δραστηρία σε θέματα βιοασφάλειας και σε ό,τι αφορά τους χημικούς φορείς και σε σχέση με τους συναδέλφους από, από το Σαχέλ που προφανώς ασχολούνται πιο πολύ με τα χημικά. Αυτό αποτυπώνει και αυτά που συμβαίνουν προσφάτως στην Συρία σε ό,τι τα χημικά όπλα. Άρα είναι μάλλον δύσκολο να περιχαρακώσουμε το πεδίο. Αλλά ο κίνδυνος ασφαλώς είναι ο εξής. Ε. Προσπαθούμε να κάνουμε αξιολογήσει για τα κράτη εταίρους και να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο χώρα. Είμαστε απόλυτα ενήμεροι ότι μα πήρε κάποιο καιρό να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε ένα εργαλείο αξιολόγηση κινδύνου, μα το επεσήμανε αυτό και το ελληνικό συνέδριο. Το εργαλείο αυτό χρεια... εφαρμόζεται λοιπόν ανά χώρα για να υπάρξει ιεράρχηση των επενδύσεων με πολύ πιο συστηματικό τρόπο, το οποίο θα μα βοηθήσει για να απαντήσω και στι ανησυχίε που εκφράσατε, να προσμετρήσουμε και τον αντίκτυπο των δράσεών μα και το πώ οργανωνόμαστε. Μαθαίνουμε, προχωρώντα, μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε επί καθημερινά. Προφανώ τα πράγματα είναι δύσκολα και σύνθετα, αλλά νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τι ε, ημέρε εστίαση, είχαμε 160 εταίρου στι Βρυξέλλε, ε, συγγνώμη, 60 εταίρους, 60 χώρε και κάποιε άλλε χώρε που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στο πρόγραμμα. Δεν κάνουμε και πολύ marketing, ξέρετε, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και περιορισμένου πόρου. Το γνωρίζουμε αυτό όχι μόνο από πλευρά προσωπικού, αλλά και από πλευρά ε, χρηματοδότηση. Μετράει και αυτό. Και επίση, δεν ανοίξαμε το κέντρο αριστεία στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Είναι ένα ολόκληρο τμήμα του κόσμου το οποίο δεν το εξετάζουμε. Παρά το γεγονό ότι και εκεί φυσικά υπάρχουν κίνδυνοι για την Ένωση. Και υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα στον Ιταλικό τμήμα τη Ασία, το οποίο δεν το έχουμε καθόλου άγγιξη σε ό,τι αφορά την ε, Δημοκρατία της Νοτιού Αφρικής, τον Ειρηνικό. Αυτά τα κομμάτια μετά αγγίξαμε καθόλου. Δεν υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να επεκταθεί αυτό το πεδίο ορισμού, αλλά θα θέλαμε να περιλάβουμε κάποιες χώρες, για παράδειγμα την Αίγυπτο. Ως τώρα αρνείται να συμμετάσχει το Καζακστάν επίσης. Έχουμε κάποιες χώρες λοιπόν τι οποίε θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικέ για την ασφαλεία μα και θα θέλαμε να τι εντάξουμε στο πρόγραμμα. Δεν έχει καταστεί αυτό δυνατόν ω τώρα, Κυρίω για περιφερειακού, θα έλεγα, λόγου. Η Μέση Ανατολή είναι αυτή που είναι. Δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω και γι' αυτό αποτελεί καλή παρατηρήση από πλευρά του Εκτικού Συνεδρίου. Κάποια από τα προγράμματα που εφαρμόζονται θα έπρεπε να τα δούμε σε πολύ εθνικό επίπεδο όπου υπάρχει εντύπωση ότι δίνουμε απάντηση σε εθνικέ ανησυχίε, αλλά σε κάποιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ξεκινάμε με τόσο χαμηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ε, συνεργασία. Για να αποφύγουμε να κινηθούμε σε τέτοιο επίπεδο, Ξεκινήσαμε με ένα νέο επίπεδο υποστήριξης προς τι χώρε, όπου εκπαιδεύουμε τους ειδικού σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του πολίτη, σε ευρωπαϊκά κέντρα για να τους στάσουμε στο επίπεδο που χρειάζονται, για να μην χρειάζονται εκπαίδευση από περιφερειακά προγράμματα. Έχουμε λοιπόν αυτό το επιπρόσθετο εργαλείο. Του φέρνουμε και στα κέντρα του ΝΑΤΟ, γιατί έχουμε και μια συμφωνία στο ΝΑΤΟ για να τους ε, ενισχύσουμε σε ό,τι αφορά την χωροφυλακή, την αστυνομία, την προστασία πολιτών, που και που και στρατιωτικούς, όταν υπάρχει σκέλος ε, προστασίας του πολίτη στις στρατιώτες, στις στρατιωτικό σκέλος, συνοριοφύλακες και του καθεξής. Όλα αυτά τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την προστασία των πολιτών στις χώρες. Προκειμένου να προσεγγίσουν τα πραγματικά περιφερειακά προγράμματα Και αυτό σχετίζεται φυσικά με το γεγονό ότι πολλέ από αυτέ τι φτώχε βρίσκονται σε ένα καθεστώ μεγάλη φτώχεια. Η πολιτική τώρα κινητοποίηση. Έχουμε εργαστεί με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση προκειμένου να προαγάγουμε τον διάλογο περί τη ασφάλεια επιτάπητο πολύ παραπάνω και μέσω των πρεσβειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρε αυτέ, στις περιφέρειες αυτέ. προκειμένου τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί χρησιμοποιούμε και τι δικέ του υπηρεσίε για να εφαρμόσουμε το project αυτό. Μία μεγάλη προτεραιότητα και στο σημείο αυτό θα διακόψω, γιατί νομίζω ότι φτάνει. Ένα καλό σχόλιο από πλευρά του Δελεκτικού Συνεδρίου, το οποίο δεν είναι και εύκολο, είναι οι χώρες εταίροι να εκπαιδεύσουν και τους άλλους με τους δικούς τους πόρους. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, στην Βορειοαφρική, στα Χέλ, η Αλγερία είναι πολύ πιο αναπτυγμένη από την το για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι υποδομέ ασφαλεία και του καθεξής. Άρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε, να πείσουμε τους Αλγερινούς να εκπαιδεύσουν τους γειτονέ τους και όχι μόνο να εκπαιδευτούν από Ευρωπαίους. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί είναι λίγο περίεργο να υπάρξει εκπαίδευση των ε, γειτόνων. Σε κάποιες περιστάσεις χρειάζεται ευρωπαϊκή δύναμη για να υπάρξει ιδιωτερότητα. Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, προχωράει η πρωτοβουλία αυτή, γιατί το πνεύμα της όλης πρωτοβουλίας φτάνει σε ένα σημείο που μπορούμε πλέον να συζητήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν είναι πάντα απλά τα πράγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τον περσικό κόλπο, για παράδειγμα. όπου οι σχέσεις μεταξύ Κατάρ και γειτόνων ασφαλώς είναι χειριστέ. αλλά υπάρχει και κέντρο αριστεία Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, ήταν στην ίδια αίθουσα. Οι εκπρόσωποι των χωρών αυτών θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν κοινά έργα. Αυτό φυσικά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές επιτυχίες οι οποίες κρύβονται πίσω από τα εκατομμύρια, από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και έχει μια κάρτα να παίξει. Θα σταματήσω εδώ και πολλά άλλα ασφαλώς ε, δεν τα ανέφερα, αλλά ευχαριστώ και πάλι το ελεκτικό συνέδριο για τη βοήθεια. Για το τμήμα του κινδύνου μπορούμε να κάτσουμε να τα συζητήσουμε το πώς θα προσμετράμε όλα αυτά. Άλλο σημείο αυτό, αλλά σημειώνουμε αυτά που μας είπατε και θα συνεχίσουμε τη βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως ε, η κυρία Γιάκοφσεν από το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ καλό το να διευρύνουμε και είναι πολύ σημαντικό η, αυτή η κουλτούρα του ελέγχου να διευρύνεται, όμως είναι αλήθεια πως θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και να εμβαθύνουμε στους ορισμούς, στους στόχους που κάθε φορά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Κύριε Γιάχοφσεν, σας δίνω λοιπόν το λόγο για να ολοκληρώσετε. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ αναγνωρίζω τα τις παρατηρήσεις. Σε τέσσερα χρόνια θα, γίνει, θα δοθεί συνέχεια σε αυτόν τον έλεγχο και τότε θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις ανάλογα με αυτά που είπε η Κομισιόν. Νομίζω πως έτσι συνοψίστηκαν πολύ καλά οι πρωτοβουλίες ε, για τις ε, ελέγχους και τις εκθέσεις. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε έτσι και πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. θα χρειαστεί οι χώρες να μπορέσουν να συνεργαστούν και να συμβιβαστούν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο σημείο 5. Έχουμε εδώ τον κύριο Παρνιό, τον εισηγητή. Είναι ο εισηγητή για την ειδική έκθεση αριθμό 15 του 2018, απαλλαγή 2018 και πρόκειται για την ενίσχυση των ε, δυνατοτήτων των δυνάμεων εσωτερική ασφάλεια στον Νίγηρα και το Μαλί. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πριν να δώσω το λόγο στον εισηγητή, να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάκοφσεν που θα μας παρουσιάσει την έκθεση ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Και μετά εσύ θα μας ε, μιλήσεις. Ναι. Κυρία Γιάκοφσεν, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε την ειδική έκθεση για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλεία στον Νίγηρα και στο Μαλί όπου είναι ομοσπονδιακά κράτη στη Δυτική Αφρική, είναι νεαρές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες με αδύναμες οικονομίες και με αναπτυσσόμενους διοικητικούς μηχανισμούς. Το Μάρτιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια στρατηγική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ με βάση ότι η ανάπτυξη και η ασφάλεια αναπτύσσονται αμοιβαία και ότι οι περιφερειακές ανάγκες χρειάζονται περιφερειακές λύσεις. Έχουμε κοινέ ε, δράσεις στρατιωτικού τύπου, αλλά και άλλα μέσα ευρωπαϊκά για να εφαρμοστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε αποστολές στον Νίγηρα και στο Μαλί για να ανταποκριθούν στις απειλέ, στην ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια τη περιοχή του Σαχέλ και στην ασφάλεια της Ένωσης. Στόχος ήταν να βελτιωθούν οι δυνατότητες των εθνικών δυνάμεων προσφέροντας κατάρτιση ε, και εξοπλισμό. 69 εκατομμύρια ευρώ για από το 2011 μέχρι το 2017 και ακόμα 66 το, για τα έτη 2014 μέχρι 2017. 69 και 66 εκατομμύρια. Εμείς θελήσαμε να δούμε πώς ε, ε, λειτουργούν οι αποστολές UCAP στο Νίγηρα και το Μαλί, αν όντως και πώς ενισχύονται οι δυνατότητες των αρχών που είναι αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια στις δύο χώρες. Ε, στέσαμε τα, ε, τα ερωτήματα του κατά πόσο ε, το σχέδιο της ΕΙΑΠ ε, λειτουργήσε ή όχι. Ε, τι βρήκαμε λοιπόν σε αυτόν τον έλεγχο. Διαπιστώσαμε ότι οι αποστολές ενίσχυσαν όντως τις δυνατότητες των αρχών για την εσωτερική, αρχή, ε, εσωτερική ασφάλεια, συγγνώμη, αλλά ότι η πρόοδο ήταν πολύ αργή και ότι υπήρχαν λειτουργικές ανεπάρκειες. Διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό της αποστολής δεν αλάμβανε επαρκή πρακτική καθοδήγηση και στην ε, περίπτωση της Γιούκα Σαχέλνη Γυράς ε, ε, δεν έλαβαν αρκετή κατάρτιση πρώτης ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων. Δόθηκε όμως τόσο στήριξη και διαδικασίες που δεν τέριαζαν στην συνθήκες εργασίας επιτόπου. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα των αποστολών επηρεαζόταν αρνητικά λόγω των διετών εντολών, ενώ είχαν ετήσιο προπολογισμό, πράγμα που δεν ενθαρρύνει τη μέσο και μακροπρόθεσμο ε, σχεδιασμό. Αν και οι αποστολές αυτές δεν, ε, δεν θέλουν να είναι μόνιμο χαρακτηριστικό των χωρών, δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου διαπιστώσαμε ότι οι αποστολές εργάζονται προς το να είναι βιώσιμες οι δραστηριότητε τους, αλλά με λιγοστή επιτυχία. Και αυτό οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της χώρες υποδοχής και εν μέρη στην ανεπαρκή συνέχεια από τις ίδιες τις αποστολές. Επίσης, οι δείκτες απόδοσης ήταν αδύναμοι και στη διάρκεια της περίοδου ελέγχου οι αποστολές δεν παρακολούθησαν και δεν αξιολόγησαν σωστά τη ε, επιτεύγματά τους. Αν και οι αποστολές είχαν παίξει σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρχών που είναι αρμόδιες για την ε, ασφάλεια στο Μαλί και στον Νίγηρα. η διαδικασία ήταν πολύ αργή και περιορισμένη. Στην έκθεση του ελέγχου ε, συστήνουμε πως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Κομισιόν θα πρέπει να βελτιώσουν την ε, λειτουργική απόδοση, να βελτιώσουν ε, τη στελέχωση, να θέσουν ε, συγκεκριμένη ε, ημερομηνία λήξης και στρατηγική εξόδου να δώσουν βελτιωμένους δείκτες για την, ε, όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση δέχτηκαν τις συστάσει μα και θέλω να του ευχαριστήσω για τη συνεργασία του. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ, κυρία Γιάκοψεν, και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Παρνιώου. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Γιάκομσεν για την πολύ συγκεκριμένη παρουσίαση που μας έκανε για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τη χρηματοδότηση των δυνατοτήτων των αρχών ασφάλειας στον Νίγηρα και στο Μαλί. Όπως το θυμήσατε κυρία Γιάκοψεν, Περισσότερο από ποτέ η περιοχή του Σαχέλ έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, άκρα φτώχεια, κρίση επιστημιστική, τρομοκρατία, συγκρούσεις, άτακτη παράνομη μετανάστευση και κλιματικότητα όπως η εμπορία ανθρώπων και διακίνηση μεταναστών. Η ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ είναι λυπής και είναι απαραίτητη για την αρμονική ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής. Γι' αυτό και είναι σημαντικό σήμερα να μπορέσουμε να δούμε αν οι δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί και στον Νίγηρα είναι ε, ε, αποτελεσματικές. Ξεκίνησαν το 12 και το 14 οι αποστολές ΕΟΚΑΠ Σαχέλ Νίγηρας και ΕΟΚΑΠ Σαχέλ Μαλί και έλαβαν 69 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και το 2017 για τον Ήγηρα και 66 εκατομμύρια ευρώ ανάμεσα στο 2014 και το 2017 για το Μαλί. Σημαντικά κονδύλια τα οποία επέτρεψαν την ενίσχυση των εσωτερικών αρχών ασφάλειας μέσα σε αυτές τις δύο χώρες. Έγινε όμως αυτό, η απάντηση είναι ναι οι εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν ενισχυθεί χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στον Νίγηρα όσο και στο Μαλί. Όμως θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες σήμερα ώστε οι δράσεις μας επιτόπου να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο μόνιμες. Στην έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο τονίζει ότι η έλλειψη επιχειρησιακών στοιχείων έχει αποτελέσει εμπόδιο επί της, μορφή, μορφής Χρειάστηκαν 18 μήνες μέχρι ότου να πάρει νομική μορφή η ΕΟΚΑ ε, δηλαδή τότε ο επικεφαλής της Απόστολης ανέλαβε προσωπικά όλες τις ευθύνες. Πώς γίνεται κανένα συγκεκριμένος ε, κονδύλι να μην έχει γρήγορα τεθεί στη διάθεση μιας τέτοιας ε, αποστολής. Ακόμα χειρότερο η ασφάλεια του προσωπικού διακυβεύθηκε όταν ε, υποχρεώθηκαν να μείνουν και να εργάζονται σε ένα ξενοδοχείο χωρίς καμία ιδιαίτερη ασφάλεια. Είναι πραγματικά απίστευτο το προσωπικό αυτό να μην έχει ε, λάβει καμία κατάρτιση και καμία βοήθεια για την εκμάθηση των διαδικασιών και των project επιτόπου. Αυτή η έλλειψη κατάρτιση σίγουρα οδήγησε σε καθυστερή στην εφαρμογή αυτών των στην υλοποίηση αυτών των αποστολών. Επίσης, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου εντοπίζει τις δυσκολίες κάλυψης των κενών θέσεων στο πλαίσιο αυτών των δύο αποστολών. Σήμερα το ποσοστό ε, κάλυψης είναι 72% στον Ήγυρα και 76% στο Μαλί. Αυτή η έλλειψη προσωπικού αποτελεί βέβαια ένα ακόμα μια τροχοπέδι ε, στην απόδοση αυτών των δύο αποστολών. Θα πρέπει γρήγορα να κάνουμε τα εξή, να προτείνουμε αποσπάσεις πιο μακροχρόνιες από το προσωπικό των κρατών μελών προς αυτές τις αποστολές. Δεύτερον, να ε, ε, προσφύγουμε στους προσωρινούς υπαλλήλους αλλά και να ε, κάνουμε κλήσεις για ενδιαφερόμενους ανθρώπους ώστε να μπορεί να επιταχυνθεί η πρόσληψη νέων ανθρώπων όταν ε, χειρεύουν οι θέσεις. Τώρα, για την ε, βιωσιμότητα αυτών των αποστολών θα πρέπει να προτείνουμε κατάρτιση ε, συμβουλές, ε, ε, υλικό, έτσι ώστε όντως αυτές οι αποστολές να είναι αποτελεσματικές. Το είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο. Αλλά δυστυχώς εκεί δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία. Η δυνατότητα διάρκειας συνδέεται με μια έλλειψη πολιτικής βούλησης και έλλειψη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αυτονομία των αρχών ασφαλείας εσωτερικά και να μην εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές αποστολές και έπειτα να εξασφαλίσουμε πιο στενή παρακολούθηση της χρήσης των καταρτήσεων που γίνονται και του υλικού που παρέχεται. Συμπέρασμα, κυρία Πρόεδρε, η κυρία Γιάκομψεν, εγώ θέλω να υπογραμμίσω πως η έκθεση του, συνεδρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου μας ε, θα να εκπονήσουμε σαφείς στρατηγικές για έξοδο για αυτές τις δυο αποστολές, ώστε να μπορέσουν, μπορέσει το προσωπικό των συγκεκριμένων αποστολών να προβλέψει και να βασίζεται συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και αυτά περιλαμβάνονται και στην έκθεσή μου που θα σας διαβιβαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Muchas gracias, señor ponente. Ah, sí. Voilà. Eh, ahora veo que el señor Seller sí tiene interés. Señor Seller. Ο κύριο Σέλερ ενδιαφέρεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και το λεκτικό συνέδριο, την κυρία Γιάκοψεν και την ομάδα τη, η οποία Μα παρουσίασαν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και λεπτομερή έκθεση και για τα πολύ σωστά σχόλια από πλευρά ε, του εισηγητού μας, του κ. Παρνιό. Η έκθεση καταδεικνύει πόσο συχνά η φιλοδοξία και η πραγματικότητα ε, απέχουν. Επενδύουμε πολλά χρήματα, αλλά τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι περιορισμένα. Μέτρια. Αυτό έχει να κάνει για μένα και με το γεγονός ότι σχεδόν όλα αυτά τα κράτη είναι σε πτώχευση. Δεν έχουν δικιά τους χρηματοδότηση, δεν έχουν δικό τους προπολογισμό και άρα εξαρτώνται από εξωτερική βοήθεια. Εκ παραλλήλου η κατάσταση της ασφάλειας είναι παραπάνω από ευάλωτη, είναι απειλητική θα έλεγα. Παράλληλα, στον Ήγηρα ότι είναι πολύ σημαντική χώρα για τις πρώτες ύλες και την παροχή πρώτων υλών σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά εργοστάσια των Γάλλων. Αλλά έχουμε πλήρη κατοχή των περιοχών αυτών από ομάδες οργανική, ε, Ισλαμικής επιρροής. Και έτσι λοιπόν οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να προβούν σε τέτοιε δράσει για να αποφύγουν τα χειρότερα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή, ότι ο συντονισμό των μέτρων μα, ε, τα πολιτικά, στρατιωτικά μέτρα συνεχίζονται και διεξαγάγονται χωρί συντονισμό εκ παραλίλου και τα κράτη-μέλη επενδύουν ε, στις περιοχές αυτές, στις χώρες αυτές, χωρίς από την απαραίτητη δικτύωση. Και όπως είπε το ελεκτικό συνέδριο και ο κ. Παρνιώτη τίθεται και το θέμα της βιωσιμότητας. Εκπαιδεύουμε δυνάμεις ασφαλείας που δεν ξέρουμε κατά πόσο στη συνέχεια θα μπορούν να πληρώνονται σωστά από το κράτος και έτσι να φροντίζουν για την ασφάλεια στις χώρες τους. Ή κατά πόσο κάπου θα χαθούν και στη συνέχεια θα απειλούν αντίθετα τους πολίτους, γιατί δεν θα πληρώνονται σωστά. Κατανοώ ότι φτιάχνουμε και καταστάσεις ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά λείπει ο απαραίτητος εξοπλισμός. Και δεν μπορεί να γίνει σωστή εκπαίδευση. Η έκθεση αυτή δεν θα απασχολήσει μόνο εμάς, αλλά και τους συναδέλφους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη χρειάζεται ε, ασφάλεια και η ασφάλεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανάπτυξη. Και χρειάζονται κυρίως κοινέ προσπάθειες, όχι στα ευρωπαϊκά θεσμικά κράτη, αλλά σε όλα τα επίπεδα για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί οι πολιτικές ε, ισορροπίε και τα καθεστώτα τα οποία αντιμετωπίζουμε δεν είναι τα ίδια με αυτά που έχουμε συνηθίσει σε δημοκρατικό επίπεδο. Διευθέτω, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθοράς και το καθεξή, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πιο καταπήγοντα παρά ποτέ στι χώρε αυτέ. Και αυτό μπορεί να έχει ω αποτέλεσμα ότι πολλοί πολίτε από τι χώρε αυτέ προσπαθούν είτε να φύγουν από τι χώρε αυτέ, είτε να αντιταχθούν και να συνασπιστούν κατά των καθεστώτων. Πολύ σύμφατα λοιπόν ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν στην έκθεση αυτή και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα πάρουμε πολύ στα σοβαρά και να τα κοιτάξουμε και στις μελλοντικές συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και το Ελληνικό Συνέδριο και τον συνάδελφο Παρνιό. Ευχαριστούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάποιος. Για το τμήμα για την Αφρική. ο σαν Λάγκ, κάπως έτσι. Εσείς, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ. Ναι, εκπροσωπώ το τμήμα διαχείρισης, ε, πολιτικής διαχείρισης των κρίσεων για τις μη στρατιωτικές αποστολές ε, στο πλαίσιο της ε, ΕΠΑ. Έχουμε εργαστεί διαμακρών με τους ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Δεχθήκαμε τις συστάσεις της έκθεσης, όπως υπόθηκε, υπογραμμίζοντας βέβαια πολλά πράγματα, όπως ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικότερο πλαίσιο στο Σαχέλ, Μαλή, γύρια. Αυτό έχει σημασία στην προσπάθεια να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των αποστολών. Στην Ιγέρια και στο Μαλή η αποστολή ήταν ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τις αστερικές ε, δυνάμεις ασφαλείας. Είναι μακρόπνες μεταρρυθμίσεις αυτές και βέβαια απαιτούν από πλευράς ε, της κυβέρνησης και των διαφόρων φορέων να αναλάβουν ε, την ευθύνη επιτόπου αυτής της ε, μεταρρύθμισης. Αν προσπαθήσουμε βράχη πρόθεσμα να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των προσπαθειών των αποστολών αυτών, μπορούμε ενδεχομένως να εκτιμήσουμε ότι ήταν μικρός. Αλλά χάρη στην παρουσία αυτών των αποστολών και τις δράσεις τους, ιδίω ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών στρατηγικού χαρακτήρα σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο στερικών ε, δυνάμεων στερική ασφαλεία. Ε, Στόχο αυτών των αποστολών ουσιαστικά η διάρκεια, η συνέχεια. Όταν μιλάμε για κατάρτιση, για εκπαίδευση, αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι παρά ένα εργαλείο μόνο στο πλαίσιο ενό συνόλου μεταρρυθμίσεων. Ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό που πρέπει να το υπογραμμίσουμε και για το οποίο εργαζόμαστε όλο και περισσότερο και με αποτελεσματικότητα θα έλεγα πλέον μαζί με τα άλλα μέσα το τμήμα των αναπτυξιακών σκέλος κομισιών με μέσα όπως είναι το καταπίστευμα επίκουσα βοήθεια για την περιοχή του Σαχέλ και με του συναδέλφους μας ε, που ασχολούνται με τα στρατιωτικά ζητήματα και το EUTM ε, για το Μαλί στρατιωτικός και άλλος των επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, οι αποστολές της ΕΠΑ είναι στα χέρια των κρατών μελών. Γίνονται αναφορές από την Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπική Ασφάλεια κάθε 6 μήνε και από το 2012 για την Ήγερα και από, από τον μάλλον και το 2014 για το Μαρίτα κράτη-μέλη ε, έχουν επανειλημμένω εκφράσει την ικανοποίησή τους για την αποτελεσματικότητα των αποστολών στον Ήγυρα και στο Μαλί. Όχι ότι είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τα τεχνικά και πολιτικά εργαλεία που υπάρχουν. Αυτά. Ευχαριστώ και αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστω να απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ζαγόν Μπουαγιόν για τον Ήγηρα από το desk. Είστε εδώ, με έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Τα είπε η επικεφαλής η μας. Ε, θέλω να πω απλά ότι ήμουν και εγώ στην αποστολή στον Νίγηρα, μία μικρή διευκρίνηση. Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει κανείς τον αντίκτυπο των ε, ε, συμβουλευτικών δραστηριοτήτων. Ε, έκαναν οι ελεγκτές ένα benchmarking και κάποιες φορές διαρωτώ με γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο χρώμα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείται μια τέτοια συμβουλευτική δραστηριότητα σε βάθος χρόνου. Δεν είναι το ίδιο με, μια, ε, με την παροχή μια κατάρτιση που ξέρουμε άμεσα αν, είχε, αν έχει επιτύχει του στόχους. Το ε, ίδιο δεν συμβαίνει με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτά είχα να πω. Μάλιστα. Θέλει κάποιος το λόγο στο τελευταίο αυτό σχόλιο, μήπως να σχολιάσει. Θέλω να πω, το ξέρω και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και οι εξωματικοί τη Κομισιόν ότι πάντοτε εμεί υπογραμμίζαμε την ανάγκη να υπάρχει συμφωνία και σύγκληση σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των δικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχουμε με το Ελεκτικό Συνέδριο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι προφανές πως δεν είναι εύκολο ούτε να δρομολογηθεί, ούτε να αξιολογηθεί ο προϋπολογισμός αυτός ε, βάσει αποτελεσμάτων, γιατί λείπουν οι δείκτες κομισιών. Πρέπει να έχετε του δικού σα δείκτε. Εντάξει, δεν είπα ότι πρέπει να συμφωνήσετε οπωσδήποτε με τους δείκτες του δείκτε του ελεγκτικού συνέδρου. Πάντω, κάποιου δείκτε πρέπει να έχετε για την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ε, και το ίδιο ισχύει και για την παροχή συμβουλών. γιατί μιλάμε για έναν προπολογισμό βάσει αποτελεσμάτων. Εντάξει, μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι αυτή η έκθεση προφανώς ε, έχει περάσει από την ε, συνήθεια διαδικασία FSA. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για τα διάφορα σχόλια. Θα το συζητούσα με χαρά σε διμερές επίπεδο, αν χρειάζονται πιο πολλές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία μας, γιατί αυτό που κάναμε ήταν να πάρουμε συνεντεύξεις από το προσωπικό, από τους εμπλεκόμενους φορείς και να αξιολογήσουμε με οποιοδήποτε το είχαμε την διαθεσιμότητα παροχής συμβουλών ορόσημων και ούτω καθεξής. Να πω ότι πρόκειται για μια έκθεση η οποία και αυτή θα ακολουθήσει την κανονική διαδικασία follow-up από πλευρά μα και ελπίζω σε 3-4 χρόνια, όταν θα επανέλθουμε, να έχουμε διαπιστώσει κάποια βελτίωση. Γιατί πρόκειται για πραγματικά σημαντικέ ε, πρωτοβουλίε και θα ήταν κρίμα σε 3-4 χρόνια να διαπιστώσουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδο. Ότι μιλάμε και για πολλά χρήματα που θα πάνε την την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Ζήλ θέλει να πάρει το λόγο. Δεν σε είδα. Ναι, πρόεδρε. Να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε και εσείς άλλωστε, το οποίο και επανέλαβε και η κυρία Γιάκοψεν, προφανώς. Τη στιγμή που θα υπάρχουν δείκτες, θα πρέπει να είναι δικοποιημένοι. από το 2012 και στον Ήγρα και στο Μαλή σε ό,τι αφορά την Υποεπιτροπή Άμυνα τη ε, Κόλπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ως Ευρωπαίος αλλά και ως Γάλλος ε, βουλευτής ε, και το έχω τονίσει αυτό και στον πρόεδρο τον Φρανσουά Ολάντ Και αυτό που είπε ο κ. Ζέλερ πριν από λίγο. Ότι η στρατιωτική παρέμβαση από πλευρά της Γαλλίας είχε τα αίτια που είχε. Και σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ευρωπαίων στην περιοχή, στέκουν αυτά που διαπίστωσε το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό όμως να προβούμε σε συστάσει προκειμένου τα πράγματα να βελτιωθούν περαιτέρω στο, μέτρο, στο μέλλον σε σχέση με τις, τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η ειδική έκθεση, όπως πάντα, ε, θα ενταχθεί στη διαδικασία απαλλαγή για το 17, οπότε θα τα ξανασυζητήσουμε. Αν δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα, δεν βλέπω. Επομένως, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ελπίζοντας και ευχόμενοι να βελτιωθεί η κατάσταση ε, στην 21η αυτή μέρα απεργίας τους. Εδώ ολοκληρώνουμε και θα τα ξαναπούμε στις 11 Ιουλίου. Γεια σας.